Okay, colleagues, can we perhaps look to uh, make a start? Uh, um, the chair, Mrs. Η κυρία Κρέσλερ, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, θα έρθει όπου να είναι από ό,τι μου είπαν, αλλά παρόλα αυτά ας ξεκινήσουμε εμείς. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Έχουμε λοιπόν την έγκριση ε, της ημερησίας διατάξεως αφού όλοι συμφωνείτε. Στο δεύτερο έχουμε ακοινήχηση της Προέδρου. Να σας πω δύο λόγια λοιπόν για το γλωσσικό καθεστώς. Ε, έχουμε λοιπόν διάφορες γλώσσες μεταξύ των οποίων τα ελληνικά ε, και επίσης έχουμε και το web streaming, τη μετάδοση μέσω ίντερνετ. Ε, τώρα ξεκινάμε η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σημείο 3, σχέση κόστος αποτελεσματικότητας του 7 προγράμματος έρευνας. Η Μαρτίνα Τζαμπαλόβα και η Νέσα Γιάλα Σέντερ είναι οι συνεισηγήτριες. Νέσα θέλεις να πεις κάτι? Όχι. Ωραία, επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε άμεσα την ψηφοφορία μας. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με την τροπολογία υπερθμών 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, 5 ελεύθερη ψήφος από ό,τι φαίνεται υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση άρχεται η ψηφοφορία Ψηφίσα... ψηφίσατε όλοι υπέρ της ψηφοφορίας 10 υπέρ 10 κατά σε αυτή την περίπτωση απερίφθη. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 8 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 11 ψήφι υπέρ, 10 κατά. 10 υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 11 ελεύθερη ψήφος υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε μια επαλήθευση και επί της τροπολογίας αυτής άρχεται πέρα της ψηφοφορίας απερίφθη 10 υπέρ 10 κατά Κάποιος πρέπει να έρθει για να αλλάξει αυτή η ισοψηφία. Τροπολογία ρυθμών 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 free votes υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται την 14 δεν την ψηφίζουμε γιατί αφορά γλωσσική τροποποίηση τροπολογία 15 Προφορική τροπολογία, συμφωνείτε όλοι με την προφορική τροπολογία. Ωραία, επομένως ε, με εντεταγμένη την προφορική τροπολογία ψηφίζουμε τη 15 υπέρ, κατά η Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 15 για μία ακόμα φορά. Πέρα της ψηφοφορίας, 11 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Σούπερ αποτέλεσμα, μπράβο. Έκανε διαφορά αυτή η μία ψήφος. Λοιπόν, τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας το ελέγξουμε και αυτό. Είναι τόσο στενό το αποτέλεσμα και κοντινό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 12 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Επομένως εγκρίνεται. 12 υπέρ, 9 κατά. Παρατηρήσει εκτό μικροφώνου οι διερμηνεί δεν ακούν προφανώ κάποιο μηχάνημα δεν λειτουργήσε. Επόμενη τροπολογία, υπαριθμό 17 υπέρ, κατά, αποχέ. απερίφθη. Τροπολογία 18, free vote υπέρ, κατά, αποχές, Ας ε, ελέγξουμε ηλεκτρονικά το αποτέλεσμα της τροπολογίας 18, πέρας της ψηφοφορίας, 11 ψήφοι υπέρ 10 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19, ελεύθερη ψήφος υπέρ κατά. Αποχές. Θέλετε να ελέγξουμε. Νομίζω θα είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Α, καλύτερα μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας της ψηφοφορίας, 11 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 20, ελεύθερη ψήφος υπέρ, κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 21 με μια προφορική τροπολογία, αντίθεση καμία ως προς την προφορική τροπολογία, επομένως τροπολογία 21 με την προφορική τροπολογία ενταγμένη υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πέντε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία υπαριθμών 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επί της παραγράφου 24 έχουμε μία προφορική τροπολογία. Συμφωνείτε όλοι με την, προφορική, με την ένταξη της προφορικής τροπολογίας. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32. Υπέρ, κατά. Αποχές προτιμώ να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία από τις τροπολογίες 32 πέρας. Απορρίπτεται 10 ψήφοι υπέρ, 10 κατά. Τροπολογία 33 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε και την 33 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 9 ψήφοι υπέρ 13 ψήφοι κατά απερίφθη τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 Θέλετε να ελέγξουμε. Ε, όχι, έκανα λάθος λέει ο Πρόεδρος. θέλω να πω ότι εγκρίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει καλύτερα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, ε, ναι, εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά. Αποχές. Απερίφθη. 45 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 46 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ή 48 δεν ψηφίζεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53 κατά τμήματα. Το πρώτο τμήμα δεν έχω το σωστό κατάλογο ψηφοφορίας λέει ο Πρόεδρος. Υπέρ του πρώτου τμήματος κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Νομίζω να κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση για το δεύτερο τμήμα. Τροπολογία 53, δεύτερο τμήμα, πέρας της ψηφοφορία. 11 ψήφοι υπέρ, 11 κατά. Απερίφθη. Τροπολογία 54, υπέρ, κατά. 54, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 55 Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 54 πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 60 υπέρ Κατά, ε, συγγνώμη, ε, πέρα της πληροφορίας, 11 ψήφοι υπέρ, 11 κατά, η τροπολογία 61 υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση και επί της τροπολογίας 61 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. Τροπολογία 62 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη τροπολογία 63 με προφορική τροπολογία Ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία διονομαστικής κλίσεως. Ονομαστική ψηφοφορία λοιπόν για το σύνολο πέρας της ψηφοφορίας. Και εδώ δεν είναι καθόλου προβληματικό το αποτέλεσμα, ούτε στενό. 22 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή εγκρίνεται λοιπόν. Yeah. So next. After the celebrations, perhaps we could... Uh, Μετά του εορτασμού μπορούμε να συνεχίσουμε με την διάταξη. Η Πρόεδρος κυρία Γκρέσλε δεν είναι ακόμα εδώ. Από ό,τι ξέρω θα ήθελε να παρευρίσκεται στις συζητήσεις για το σημείο 4, για την αντιπροσωπεία, την αποστολή στην ε, Ουάσιγκτον, της οποίας ε, θα προεδρεύσει. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 5. Είναι εδώ το ελεγκτικό συνέδριο. Ωραία και ο εισηγητή τη Έκθεση, οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Απαιτούνται περισσότερε προσπάθειε για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του. Δόκτω, πώ μπορείτε να συνεχίσετε, να ξεκινήσετε τη συζήτηση ω εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρίε και κύριοι, επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω το ελληνικό Συνέδριο για την έκθεση που έχει καταρτήσει. Γιατί η έκθεση αυτή για πολλούς λόγους είναι ιδιαίτερως ε, σημαντική. Πρώτα απ' όλα έχουμε το πρόγραμμα Natura 2000 και τους ε, πόρους ε, που έχουν αφοσιωθεί στα Natura 2000 και δεύτερον είναι σημαντικό να καταδείξουμε ότι αυτή η έκθεση είναι μια ειδική έκθεση που ε, θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο αυτό το πρόγραμμα. Να περιμένω μήπω ε, να επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα. Συνάδελφοι, παρακαλώ ησυχία για να ακούσουμε όλοι τον εισηγητή. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια ειδική έκθεση λοιπόν του Ελεκτικού Συνεδρίου που εξετάζει το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα της ε, φύσης. Και δηλώνω την απογοήτευσή μου από ε, τον έλεγχο. Τα συμπεράσματα δηλαδή της έκθεσης, γιατί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ε, πρωτοπόρο ε, σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντο. Όμω υπάρχουν ε, πολλά προβλήματα, πολλέ αδυναμίες. Η προστασία τη βιοπικιλότητα, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα και τι πιο σημαντικέ προκλήσει. Η στρατηγική 2000 που θα πρέπει να ασχοληθεί ακριβώ με την προστασία και τη διατήρηση τη βιοπικιλότητα στα κράτη-μέλη, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο. Τα κράτη-μέλη δεν δίνουν αρκετή έμφαση, δεν καταβάλουν επαρκείς προσπάθειες προκειμένου αυτή η στρατηγική να μπορέσει να αξιοποιηθεί πλήρως ε, με βάση την ε, εφαρμογή της και να δούμε ποιε ε, είναι οι βελτιώσει που μπορούμε να επιφέρουμε στη στρατηγική. Με εξέπληξαν δύο στοιχεία. Αφενός, Ε, η φύση δεν γνωρίζει σύνορα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συντονισμό μεταξύ κρατών μελών. Όμω, ο συντονισμό και η συνεργασία μεταξύ κρατών μελών σε ό,τι αφορά την προστασία τη βιοποικιλότητας δεν λειτουργεί σωστά. Μετά, τα διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη που ε, παρεμβαίνουν ε, ούτε αυτοί πληρούν και επιτελούν τον ρόλο του. Δεν υπάρχει σαφή και επαρκή ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να δούμε πώς πήγε η εφαρμογή της στρατηγικής Natura 2000. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να έχουμε έγγραφα, πληροφορίε, στοιχεία που θα είναι μάλιστα στοιχεία σαφή και ακριβή και θα απευθύνονται προ τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό ε, συνιστώ τα κράτη-μέλη να είναι σε θέση να αξιολογήσουν την πρόσβασή τους σε αυτή τη διασυνορική συνεργασία και τα ενδιαφέρονα μέρη να μπορούν επίση να βελτιώσουν τους διάβλους επικοινωνίας για να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των επιμέρους μερών. Είναι πολύ σημαντικό επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει στα κράτη-μέλη, να υποβάλει μάλλον στα κράτη-μέλη στοιχεία ε, εμπειρογνωμόνων, εκθέσεις, προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους μας ό,τι αφορά την ε, διατήρηση και την επίτευξη των στόχων ε, ε, που έχουμε θέσει προγραμματικά. Υπάρχει και ένα πλαίσιο ε, προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί ως στόχοι για το Natura 2000 και όπως ανέφερα ήδη, τα κράτη-μέλη δεν έχουν δώσει αξιόπιστα στοιχεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν από εδώ και στο εξή να βρει έναν τρόπο να έχει πιο ε, αυστηρή απέτηση απέναντι στα κράτη-μέλη που δεν δίνουν ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία σε ό,τι αφορά τους τόπου Natura 2000. Και τέλο, κύριε και κύριοι, επιτρέψτε μου να κάνω ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα πρέπει όντω να καταβάλουμε επιπρόσθετε προσπάθειε ό,τι αφορά τη διατήρηση τη βιοπικιλότητα και στον τομέα τη συνεργασία μεταξύ κράτων μελών. Δεν ε, πρέπει να περιοριστούν αυτές οι προσπάθειες γιατί αν δεν τα καταφέρουμε όλες οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε δημοσιονομικό επίπεδο για το Natura 2000 θα είναι ε, απλές γραπτές συστάσεις ε, και ενώ γράμμα και δεν θα μας οδηγήσουν σε πραγματικά αποτελέσματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που έτσι δεν θα είναι σε θέση ε, να προστατεύσει αυτά που είναι, είναι πλέον πολύτιμα, δηλαδή η φύση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μπελίνες, κύριε Μιλιώνη μάλλον από το ελεγκτικό συνέδριο, αν μπορείτε να μας παρουσιάσετε την ειδική σας έκθεση. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να σας ε, παρουσιάσω την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου για το δίκτυο Natura 2000. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζετσόφσκι για τις ε, εξαιρετικά χρήσιμες συστάσεις του. Το δίκτυο Natura 2000 που δημιουργήθηκε υπό τις οδηγίες περί και οικοσυστημάτων είναι βασικό στοιχείο της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 για να περιορίσουμε και να σταματήσουμε την απώλεια βιοποικιλότητας που είναι από τις μεγαλύτερες προκλήσεις ε, στον τομέα του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο του 2000 ε, έχει πάνω από 27.000 ε, τόπους σε όλη την Ευρώπη, σημεία δηλαδή Natura 2000 και καλύπτει πάνω από το 18% Τη ε, επικράτεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και περίπου 6% της θαλάσσια ε, επικράτειας. Τα κάθε μελη είναι υπεύθυνα για την ε, διαμόρφωση, διαχείριση και χρηματοδότηση του δικτύου. Εντός έξι ετών από τον προσδιορισμό ενός τόπου ως χώρου ιδιαίτερη σημασία για την κοινότητα θα πρέπει να υιοθετηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα ε, διατήρησης ε, για να ε, αποκαταστήσουμε τα προστατευόμενα είδη και οικοσυστήματα. Δεν απαγορεύονται οι κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες στους τόπους Natura 2000, όμως τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι δεν υποβαθμίζονται έτσι αυτές οι περιοχές. Επομένως, οποιοδήποτε σχέδιο, έργο έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μια περιοχή Natura 2000 θα πρέπει να αξιολογηθεί για να δούμε ποιες είναι επιπτώσει ε, για την περιοχή. Μπορούν και οι αρμόδιες αρχές να συμφωνήσουν για ένα έργο, αρκεί τα μέτρα μετριασμού για την... Ε, έχουν προβλεφθεί αντίστοιχα μέτρα, λοιπόν, για να μετριάσουμε τον αρνητικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προσέγγισή μας για τον έλεγχο, θεωρήσαμε, εξετάσαμε μάλλον, κατά πόσο το δίκτυο έχει τύχει ε, τη κατάλληλη διαχείρισης, χρηματοδότησης και παρακολούθησης. Επισκεφθήκαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέντε κράτη-μέλη ε, με οχτώ δύο γεωγραφικές περιοχές και 24 περιοχές το 2000. Επίσης, κάναμε και μία μελέτη στα υπόλοιπα 23 κρατημέλη για να δούμε, να έχουμε ε, πληροφορίες για τα συστήματα διαχείρισής τους και την δημόσια χρηματοδότηση που χρησιμοποιήθηκε για αυτές τις περιοχές. Το βασικό μήνυμα της έκθεσής μας είναι ότι ε, ενώ το Natura 2000 διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την προστασία της βιοποικιλότητας, παρόλα αυτά απαιτείται σημαντική πρόοδος αν θέλουμε να πετύχουμε τους φιλόδοξους μας στόχους η έκθεση αναφέρει αυτό το μήνυμα σε τρία μέρη, τα οποία και εγώ αυτή τη στιγμή θα σας επισημάνω. Στο πρώτο τμήμα της έκθεσης εξετάσαμε πώς τα κράτη-μέλη διαχειρίστηκαν το δίκτυο 2000, Natura 2000. Η εφαρμογή του προγράμματος Natura 2000 απαιτεί ε, στενό συντονισμό ε, μεταξύ διαφόρων αρμοδιών αρχών στον περιβαλλοντικό, γεωργικό, βιομηχανικό και σε άλλους κλάδους και με πολλά ενδιαφερμένα μέρη, πιο συγκεκριμένα ε, τους ε, ιδιοκτήτες και χρήστες γης. Στα κράτη-μέλη βρήκαμε παραδείγματα επαρκούς συντονισμού και εμπλοκής των βασικών ενδιαφερμένων μερών. Επιπλέον, η διασυνορική συνεργασία για την προστασία κοινών ειδών και οικοσυστημάτων είδαμε ότι δεν είχε αναπτυχθεί επαρκώς τα μέτρα διατήρησης που είναι απαραίτητα για να διατηρήσουμε ή να αποκαταστήσουμε ε, οικοσυστήματα σε ό,τι αφορά την χλωρίδα και την πανίδα θα πρέπει να ληφθούν ε, επαρκώς και θα πρέπει να τους δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο για να εφαρμοστούν ε, αποτελεσματικά θεωρήσαμε ότι, και βρήκαμε μάλλον ότι υπήρξαν σημαντικές καθυστερήσεις στην υιοθέτηση αυτών των μέτρων συντήρησης και στα πέντε κρατημέλη που επισκεφθήκαμε και είχαμε παραδείγματα μέτρων ε, διατήρησης που δεν είχαν προσδιοριστεί επαρκώς ε, και έλειπαν ε, συγκεκριμένα μάλιστα για την επίτευξή τους. Σε ό,τι αφορά τώρα τα επερχόμενα σχέδια του, στις περιοχές Natura 2000, θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε υπό το φως αυτών των ε, στόχων. Σε όλα τα κράτη-μέλη ε, είδαμε ότι κάνατε τις εξολογήσεις, αλλά σε όλες τις, περι... περιπτώσεις βρήκαμε προβλήματα. Έλλειψη ανάλυσης του αντικτύπου σε ό,τι αφορά το έργο, σε όλα τα είδη και οικοσυστήματα, ανεπαρκής ε, τεκμηρίωση ή εξολογήσεις που δεν είχαν γίνει από κατάλληλα εκπαιδευμένο και επιστοποιημένο ε, προσωπικό. Ο σορευτικός αντίκτυπος ε, διαφόρων ε, έργων στις περιοχές αυτές δεν είχε ληφθεί υπόψη επαρκώ. Τέλος, η πρακτική εφαρμογή των μέτρων μετριασμού δεν ε, ελέγχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις από τις αρμόδιες αρχές. Θεωρήσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εποπτεύει την υλοποίηση του Natura 2000, όμως συστήνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει ε, τις προσπάθειές της ε, για να διαδώσει ε, τα έγγραφα καθοδήγησής της και τα αποτελέσματα των βιογεωγραφικών της σεμιναρίων. Στο δεύτερο τμήμα της έκθεσης εξετάσαμε κατά πόσο το δίκτυο Natura 2000 έχει χρηματοδοτηθεί καταλήλως. Η προσέγγιση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την χρηματοδότηση της εφαρμογής του δικτύου Natura 2000 ήταν η αξιοποίηση υφιστάμενων ευρωπαϊκών πόρων, κυρίως από την κοινή γεωργική πολιτική και από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα ταμεία συνοχής. Οι ευκαιρίε για την στήριξη του Νατούρου 2000 υφίστανται στο πλαίσιο τη στήριξη προ τη βιοπικιλότητα σε διάφορα κλαδικά ε, προγράμματα χρηματοδότηση. Ε, βρήκαμε όμως, διαπιστώσαμε, ότι δεν είχαν κινητοποιηθεί επαρκή πόροι για τη στήριξη τη διαχείριση του δικτύου Νατούρου 2000. Επίσης, δεν υπήρχαν αξιόπιστε πληροφορίε για το κόστο του δικτύου ε, και για τη χρηματοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. τα λεγόμενα PAPS, τα πλαίσια ε, προτεραιοτήτων, είναι ένα μέσο στρατηγικού σχεδιασμού που προσδιορίζει ανάγκες χρηματοδότηση και προτεραιότητε, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Έχουν εξελιχθεί και διαμορφωθεί από τα κράτη-μέλη με τη στήριξη τη Επιτροπής. Όμως, διαπιστώσαμε ότι αυτά τα πλαίσια δεν δίνουν μια πλήρη εικόνα ε, της πραγματικής χρηματοδότησης μέχρι το 2013 και ε, των ε, προβλεπόμενων πόρων που θα διοχετευθούν κατά την περίοδο 2014-2020. Το Ορατήριο 2000 ήταν μόνο ένας από τους πολλούς στόχους στα αναπτυξιακά προγράμματα που είχαν υποβληθεί από τα κράτη-μέλη για την ε, τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Και διαπιστώσαμε ότι τα έγγραφα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν τις ε, ανάγκες χρηματοδότησης που έχουμε βρει στα πλαίσια δράσης προτεραιοτήτων ε, και για παράδειγμα βρήκαμε περιπτώσεις προγραμμάτων που έχουν χρηματοδοτηθεί και καλύπτουν μόνο συγκεκριμένα ήδη και εκποσυστήματα ενδιαφέροντος ή που δεν καλύπτουν πλήρως ε, τις οικονομικές ζημίες που ε, προκύπτουν από την συμμόρφωση με τις απαιτήσει Natura 2000. Στο τρίτο μέρος τώρα της, ε, της έκθεσης εξετάσαμε κατά πόσο το δίκτυο έχει τύχη της κατάλληλης παρακολούθησης. Η παρακολούθηση και τα συστήματα παρακολούθησης και υποβολή εκθέσεων για το Natura 2000 δεν ήταν επαρκή για να παράσχουν πλήρη στοιχεία ε, για την αποτελεσματικότητα του δικτύου. Υπάρχουν δείκτες και σε επίπεδο χρηματοδότηση προγραμμάτων, όμως δεν μπορούσαν να οματοποιηθούν για να μας δώσουν μια πλήρη εικόνα των αποδόσεων σε ό,τι αφορά το δίκτυο Natura 2000 ε, και συνδέονταν με γενικούς στόχους βιοποικιλότητας και όχι με τους ειδικού στόχους των προστατευόμενων περιοχών και έδιναν έμφαση ε, στα αποτελέσματα ε, πιο πολύ τα στατιστικά και όχι στα αποτελέσματα πραγματικά στο φορά τη συντήρηση του, ε, της περιοχής. Ε, σε επίπεδο περιοχών Natura 2000 βρήκαμε ότι τα σχέδια χρηματοδότησης δεν είχαν τύχει της κατάλληλης προετοιμασίας και δεν ήταν αρκετά λεπτομερή και δεν έδιναν ιδιαίτερη έμφαση στο χρόνο, στη χρονική διάσταση. και επίσης πολλές φορές δεν ήταν επικαιροποιημένα τα, τα δεδομένα. Σε ό,τι αφορά ε, το καθεστώς ε, συντήρησης ε, πολλές φορές ήταν ελλειπή τα στοιχεία και δεν μπορούσαμε να πετύχουμε την συγκρισιμότητα. Τέλος, κάναμε ορισμένε συστάσεις για την βελτίωση της διαχείριση του δικτύου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καθοδηγήσει τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την εκτίμηση με αξιόπιστο και εναρμονισμένο ε, τρόπο σε ό,τι αφορά την στήριξη προς το Natura 2000 και να έχει κοινού ε, δείκτες για όλα τα ευρωπαϊκά ταμεία και τους ευρωπαϊκούς πόρους. Τα κάτι μέλη θα πρέπει να ολοκληρώσουν ε, την θέσπιση των, και ε, υιοθέτηση των απαραίτητων μέτρων διατήρησης, να προτείνουν μέτρα τα οποία αφορούν τις ειδικέ ανάγκες των περιοχών, να προετοιμάσουν σχέδια παρακολούθησης και να τα υλοποιήσουν. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και τώρα θα ήθελα να δώσω το ε, λόγο στα ε, μέλη αλλά και στην Επιτροπή ε, και στη συνέχεια θα επιστρέψουμε και πάλι στον γνωμοθότη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μέλος, τον κύριο Αλή. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Τζοκόφσκι, κύριε Μιλιώνη. Αρχικά ε, θα ήθελα να ε, χαιρετήσω την αναφορά από την πλευρά ε, του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου σχετικά με το δικτύο Natura 2000 όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση αλλά και, την παρακολούθηση του Νατάρου 2000 ε, ποιες ε, δραστηριότητες αφορούν την Κομισιόν και ποιες τα κράτη-μέλη. Θα ήθελε επίσης να συγχαρώ τον γνωμοδότη για την έκθεση. Έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά και καλύπτει όλες τις πλευρές ε, οι προτάσεις του για την ε, συμπερίληψη ε, στην αναφορά απολογών της Κομισιόν για το 2016 χρειάζεται βελτίωση όσον αφορά την εφαρμογή του Natura 2000. Το Natura 2000 το δίκτυο αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην προστασία της βιοπικιλότητας τόσο στην Ευρώπη όσο και, στην και η διαχείρισή της θα πρέπει να εφαρμοστεί με έναν ορθό τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν η συμμετοχή περιοχή ιδιοκτητών ε, γεών, καθώς βρίσκεται και μερών, ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο ε, και όμως υπάρχουν ε, ζητήματα τα οποία προκαλούν ε, ανησυχία ε, διότι το πλαίσιο δράσης προτεραιότητας αφορά το κόστος το οποίο παρουσιάστηκε από τα κράτη-μέλη και οι οικονομικές κατανομές για το Natura 2000 δεν, θα, δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν παρκώς και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αναφερθώ στους εκπροσώπους της Κομισιόν ε, με κάποια ερωτήματα. Η ε, επεξήγηση της Κομισιόν για ποιο λόγο ε, δεν είχε ολοκληρωθεί μέχρι το Σεπτεμβρίου του 2016 η αναφορά δεν μας έχει πείσει ιδιαίτερος. Για να μην πω κάτι άλλο. Ε, η Κομισιόν αποδέχεται την ε, πρόταση ε, να συνεχιστεί η διανομή των πληροφοριών, όμως ισχυρίζεται ότι υπάρχουν οικονομικά εμπόδια για να ξεπεραστούν, οικονομικές δυσκολίες για να περαστούν τα γλωσσικά εμπόδια και δεν νομίζω ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να μεταφράσουν από μία τουλάχιστον από τις γλώσσες που χρησιμοποιείται και από το Κοινοβούλιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν είναι σοβαρή δικαιολογία αυτή. Επίσης η Κομισιόν αποδέχεται όλες τις προτάσεις προς τα κράτη-μέλη. Μπορείτε λοιπόν να μας εξηγήσετε συντόμως ποιος μηχανισμός χρησιμοποιείται για να ε, γίνει η εφαρμογή όλων αυτών των προτάσεων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάνναγκαν, ο επόμενο ομιλητή, Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε για την έκθεση και για την ε, δουλειά του γνωμοδότη. Ε, μπορούμε να πούμε ότι ε, αν δεν υπήρχε το Natura 2000 ε, τότε εγώ δεν θα βρισκόμουν εδώ ανάμεσά σας και ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι διότι ασχολήθηκα με την ευρωπαϊκή πολιτική διότι στην Ιρλανδία είχαμε ένα περιστατικό όπου είχαμε αποφάσεις από πάνω προς τα κάτω που μας επιβλήθηκαν χωρίς να ερωτηθούμε ε, έτσι το βλέπουμε εμείς ε, και ε, όταν πολλοί γειτονέ μου άκουσαν το Natura 2000 ήταν επειδή η αστυνομία απειλούσε να τους συλλάβει επειδή χρησιμοποιούσαν καύσιμα και πιστεύουν, πολλοί πίστευαν ότι είναι ο σωστό τρόπο για να το κάνουν αυτό διότι το κάναμε και εκατοντάδες χρόνια όμως έτσι θερμαίνουμε εμείς τα σπίτια μας και τώρα ε, θα, μιλήσω, θα μιλούσα με αγγλική ή ε, βρετανική ε, προφορά διότι ο πατέρας μου θα έκανε την απόλυτη αμαρτία κάνοντας κάτι τέτοιο. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι, ε, αντιμετωπι... ότι κινδυνεύαμε με μισό εκατομμύριο πρόστιμο, ακόμα και φυλάκιση, μεγαλύτερη από ό,τι σου επιβάλλεται σε περίπτωση βιωσμό για κάτι το οποίο κάνουμε εδώ και αιώνε. Μπορούμε να συζητήσουμε για το αν είναι σωστό ή λάθο, όμω ε, δεν προσπαθώ να σας πω πώς θα λειτουργήσει καλύτερα ή όχι. Θα λειτουργούσε καλύτερα λοιπόν αν είχαν ερωτηθεί οι πολίτες εκ των προτέρων και κάτι τέτοιο δεν συνέβη ε, Πιστεύω ότι μπορούμε να μάθουμε από όλο αυτό. Είχαμε εκατοντάδες ανθρώπους ε, οι οποίοι ε, είχαν να αντιμετωπίσουν ε, την αστυνομία, δυνάμεις της αστυνομίας, οι οποίοι κρατούσαν όπλα και προσπαθούσαν να σταματήσουν τους ανθρώπους από να χρησιμοποιήσουν τη γη τους. Το αν είναι σωστό ή λάθος όλο αυτό είναι κάτι που χρήζει συζήτηση. Όμως είναι δύσκολο όλο αυτό, κατάγομαι από την Ιρλανδία που το πρώτο πράγμα που σκέφτονται οι άνθρωποι είναι ότι είναι καταπράσινη και είναι πράσινη για ένα λόγο. Διότι δεν μας αρέσει να καταστρέφουμε τη χώρα μας, τη φροντίζουμε ε, και αν είχαμε μιλήσει εκ των προτέρων για όλο αυτό σίγουρα θα είχαμε βρει μια καλύτερη λύση. Και ε, ξέρω ότι στόχος ήταν η προστασία του περιβάλλοντος και για πολύ καιρό ε, στην ε, Ιρλανδία ήταν βρώμικη λέξη ο περιβαντολόγος ε, διότι χωρίς το περιβάλλον μας δεν θα, δεν θα υπήρχαμε. Αν λοιπόν θέλουμε να γίνει όλο αυτό σωστά στο μέλλον, θα πρέπει να μιλήσουμε με τους ανθρώπους κατά τόπους, διότι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να υπάρξει ε, συζήτηση. Ε, δεν γίνεται δηλαδή να λαμβάνουμε μέτρα και στη συνέχεια ε, να γίνεται συζήτηση, διότι αυτό προκαλεί προβλήματα. Κάτι ακόμα, η αριστερά και η δεξιά δεν γνωρίζουν ε, τι ε, κάνουν. Έχουμε μια κατάσταση στην Ιρλανδία όπου έχουμε δύο πλευρές. Ε, έχουμε το Λακτάλτ, το οποίο πριν από τέσσερα χρόνια η κοινότητα της περιοχής συζήτησε επανειλημμένως ότι δεν χρειαζόταν άδεια εξόριξης και ανακάλυψαν από την οδηγία, ε, για το, ε, οδηγία πλαίσιο για το νερό ε, ότι μπορούσαν κανονικά να πιούν το νερό αλλά αργότερα ανακάλυψαν ότι υπήρχαν βλαβερές ουσίες σε αυτό. Και τελικά συνειδητοποίησαν ότι μπορούν να το πιούν μονάχα σε περίπτωση που υποστεί επεξεργασία τους είπαν επίσης ότι ε, δεν μπορούν να χτίσουν ένα εργοστάσιο επεξεργασίας νερού εκεί πέρα. Με αποτέλεσμα το, ε, οι πολίτες εκεί πέρα ή ε, θα ακολουθήσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία ή θα δηλητηριαστούν, όπου δύο νομοθεσίες αντικρούουν η μία την άλλη είναι διατεθειμένοι να μεταβούν σε μια άλλη λίμνη, είναι μια προσωρινή όμως λύση και υπάρχουν τεράστιες ε, δυνατότητες. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια κατάσταση όμως στην Ιρλανδία όπου έχουμε μια υπηρεσία για το περιβάλλον η οποία αποτρέπει τους ανθρώπους ε, να επεξεργαστούν το νερό ενώ η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ισχυρίζεται ότι δεν μπορούν να πιούν το νερό παρά μόνο άμα επεξεργαστούν το νερό. Ναι, θέλω να πιω το νερό, θέλω να προστατεύσω ε, το περιβάλλον. Έχω παιδιά τα οποία θέλω να έχουν επαφή με το ε, περιβάλλον, όμως θα πρέπει να γνωρίσουμε τι κάνουν οι δύο πλευρές μας, διότι το αποτέλεσμα είναι ότι οι άνθρωποι σε αυτή την περιοχή αντιμετωπίζουν τους ε, περιβαλλοντιστές ως τον εχθρό. Αυτό δεν είναι σωστό, όμως συμβαίνει για ένα λόγο και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Και ο ένας από αυτούς τους λόγους είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα το ερώτημα είναι πώς θα επιληθεί μας λένε να πάμε σε αυτή την περιοχή ε, και ε, λένε ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να περιμενουν τρια 3-4 χρόνια μέχρι ότου να έχουν καθαρό πόσιμο νερό. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα λοιπόν όπου σε περίπτωση που έχουμε ε, ε, διαμάχες, θα υπάρχει δυνατότητα επίλυσης και σε περίπτωση που έχουμε την υποστήριξη των πολιτών για κάτι θα συμβεί πολύ καλύτερα από ότι αν πρέπει να τους το επιβάλλουμε δεν πρόκειται ποτέ να έχει πραγματικά αποτελέσματα. Η λύση λοιπόν για όλο αυτό είναι να μιλήσετε αρχικά στους ανθρώπους και να μην υποκρίνεστε ότι και καλά θα το κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ όσον αφορά το ε, ερώτημα της ε, στρατηγικής για την ε, βιοπικιλότητα και το κατά πόσο εφαρμόζεται, εκεί υπάρχει ένα έλλειμμα και αυτό το έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει και υπήρξε μια πάρα πολύ καλή έκθεση του Κοινοβουλίου και αυτό το οποίο συζητήσαμε τότε επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έκθεση. Τους τελευταίους ε, μήνες αντιμετωπίσαμε επίσης ε, και το γεγονός ότι ε, με την καλύτερη νομοθέτηση εν τέλει έχουμε τις δύο, τους δύο πυλώνες του Νατούρο που είναι η προστασία των πτηνών και η κατευθυντήρια ΠΑΦ όλα αυτά δείχνουν ότι ε, υπήρξε μια έλλειψη ικανοποίηση από την πλευρά των κρατών μελών και είμαστε ευγνώμονε για το γεγονό ότι η Κομισιόν στην αξιολόγησή της καταλήγει ότι αυτό το οποίο επιβεβαιώνει αυτό το οποίο επαναλαμβάνουμε εμείς στο Κοινοβούλιο, το ότι έχουμε αυτές τις δύο ε, οδηγίε και το πώς θα πρέπει να εφαρμοστούν, ε, πού θα πρέπει ε, να γίνουν σχέδια αξιολόγηση, τα οποία δεν θα υπάρχουν μονάχα στο χαρτί, ότι θα πρέπει να υπάρχει η χρηματοδότηση, η νομοθεσία αυτή λοιπόν συνεισφέρει ούτως ώστε η βιοπικιλότητα όχι μόνο να αποτρέπει την απώλεια βιοπικιλότητας αλλά να συνεισφέρει ταυτόχρονα ούτως ώστε η βιοπικιλότητα να προστατεύεται και να προωθείται στην Ευρώπη. Επίσης η έκθεση ε, αναφέρει αρκετά σημεία ε, και θα ήθελα να, συνα... να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τόμος ε, για τα όσα ανέφερε και είμαι σίγουρη ότι η Κομισιόν σήμερα θα πάρει ε, πρώτη το λόγο ε, διότι με αυτή την εξαμηνία καθυστέρηση επιτέλους μας έδωσε ένα σχέδιο δράσης στις 17 Απριλίου όπου στην 27 Απριλίου όπου υπάρχει αμφιβολία σχετικά με τις επενδύσεις και να υπάρξει μια βελτίωση ε, κάτι το οποίο αναφέρθηκε από τους προηγούμενους ομιλητές. Όλα περιλαμβάνονται στην έκθεση. Ε, δεν ξέρω όμως αν για όλο αυτό θα, πρέπει, θα θελήσει να πει κάτι η Κομισιόν. Είχα τη δυνατότητα να μελετήσω εις βάθος την έκθεση ε, και ε, χαίρομαι που περιλαμβάνονται όλα αυτά ε, στην έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Όμως υπήρξε από την πλευρά της Κομισιόν μια καθυστέρηση. Ε, έχουμε όμως καλά μέσα, τα οποία όμως θα φέρουν κάποια αποτελέσματα, όμως λείπουν κάποιοι δείκτες. Ελπίζω λοιπόν ότι όλοι αυτά θα συμπεριληφθούν ε, και ε, είμαι πεπισμένη ότι όσον αφορά τους, ε, τις επενδύσεις θα βλέποντας ε, το σχέδιο δράσης ε, προβλέπονται ε, επιπλέον οικονομικά μέσα όσον αφορά την κατανομή της, του προϋπολογισμού για την κοινή γεωργική πολιτική αλλά και το 10% για την βελτίωση όχι του προϋπολογισμού live αλλά αυτό είναι ένα πολύ μικρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση όμως η Κομισιόν ίσως θα μπορούσε ε, να εμβαθύνει πάνω σε όλο αυτό το σχέδιο ε, δράσης ε, το οποίο περιλαμβάνει τα 15 βήματα. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Γιαβόρ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο ε, για την δράση του γενικότερα και για την έκθεση αυτή ειδικότερα. Μπορώ να συμφωνήσω με προραλήσεντες συναδέλφους ότι αυτό το δίκτυο Natura 2000 είναι ένα από τα σημαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ε, και μάλιστα ε, πριν από κάποια χρόνια ε, είχαμε μετά από μία σχετική μελέτη το συμπέρασμα ήταν ότι αν έχουμε κάποια πρόοδο περιβαλλοντική στην Ευρώπη ακριβώς αυτό οφείλεται στις οδηγίες που σχετίζονται με την Natura. Χαίρομαι που έχουμε την ειδική έκθεση της, του ελεγκτικού συνεδρίου για το θέμα αυτό. Ίσως πιο χρήσιμο θα ήταν αν ε, μπορούσαμε να έχουμε την έκθεση αυτή στη διάρκεια της ε, ε, διαδικασίας συζήτησης και μεταρρύθμισης της, των οδηγιών για τα πουλιά και τα ενδιατήματα. Εν πάση περιπτώσει ε, το γενικό συμπέρασμα είναι ότι είναι καλές οι οδηγίες αλλά ότι χρειάζεται βελτίωση ε, και άλλωστε υπάρχει και ένα σχετικό σχέδιο δράσης το οποίο έχει ανακοινωθεί. Ε, αλλά βεβαίως καλό θα ήταν να υπάρχει καλύτερη, καλύτερος συντονισμός ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη. Εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω κάποια από τα συμπεράσματα αυτής της ειδική έκθεσης. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό που αναφέρεται ότι τα κράτη-μέλη διαχειρίζονται αρκετά ικανοποιητικά ε, το δίκτυο Natura. Ε, ε, είναι κάτι το οποίο τα κράτη-μέλη και κάποιοι σχετικοί ευρωπαϊκοί οργανισμοί και υπηρεσίες θα πρέπει να το λάβουν υπόψη ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Ο συντονισμός επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ε, ζήτημα. Ε, το δίκτυο δεν αφορά μονάχα θέματα τα οποία άπτονται της συντήρησης, ε, αλλά υπάρχουν και άλλα υποκείμενα ζητήματα τα οποία αφορούν την ανάπτυξη της υπαίθρου κτλ. Επίσης, στην έκθεση αναφέρονται τα ε, μέτρα συντήρησης τα οποία συχνά αργοπορούν, καθυστερούν, δεν γίνονται έγκαιρα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιπροσθέτω σε ένα σημαντικό θέμα και νομίζω ότι όλοι έχουμε ε, μια μακρά σειρά ε, από προγράμματα τα οποία δεν έχουν σωστά αξιολογηθεί. Δεν αξιολογούνται λοιπόν ικανοποιητικά τα προγράμματα σε σχέση με τον αντίκτυπο που θα έχουν ε, πολλές φορές δηλαδή δίνεται πράσινο φως σε κάποια projects τα οποία μπορεί να έχουν πολύ ισχυρό αντίκτυπο ε, στο περιβάλλον ε, και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγγνώμη, νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και διάφορες υπηρεσίες ευρωπαϊκές δεν κάνουν όσα θα έπρεπε να κάνουν. Επίσης χρηματοδότηση και τρόπος ε, χρήσης ε, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Και εδώ υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν είναι απολύτως ικανοποιητικά. Πρώτον πρέπει να πούμε την πρώτη διαπίστωση ότι δεν κινητοποιούνται αρκετά ικανοποιητικά τα κονδύλια. Ε, δηλαδή μερικές φορές υπάρχει καλή προσέγγιση από τα κράτη-μέλη, μερικές φορές τα προγράμματα είναι αρκετά καλά αλλά δεν κινητοποιούνται αρκετά ικανοποιητικά τα κονδύλια κονδύλια. Επομένως θα πρέπει και ο σχεδιασμός να είναι καλύτερος αλλά και να είναι και αρκετή η χρηματοδότηση έτσι ώστε πραγματικά να μπορέσει να υλοποιηθεί η προστασία του περιβάλλοντος. Έχω και κάποιες ε, ερωτήσεις. Δυστυχώς ε, πρέπει να πω προς την Κομισιόν περισσότερο και όχι προς, τόσο πολύ προς το ελεγκτικό συνέδριο. Πρώτη ερώτηση σχετικά με την υλοποίηση και την διαχείριση ε, των ε, ε, θέσεων Natura 2000. Ρωτώ λοιπόν την Κομισιόν. Δεν είναι πολύ σαφές από το σχέδιο δράσης ότι στηρίζεται πραγματικά τα κράτη-μέλη, κυρίως δε τις περιφέρειες και τους τοπικούς εμπλεκόμενους περίπου 50% των ε, θέσεων ε, Natura 2000 έχουν ε, σχέδια διαχείρισης και πέρα από το τι περιλαμβάνει, τι είναι αυτό το σχέδιο διαχείρισης, καλό ή κακό, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο διαχείρισης, management plan και αυτό θα πρέπει να το τονίζει η Κομισιόν και να πιέζει τους εμπλεκόμενους να προετοιμάζουν ένα τέτοιο σχέδιο διαχείρισης. Προκύπτει από αυτή την ερώτηση και άλλη μία. Ε, πώς γίνονται οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη-μέλη. Γιατί η προστασία των θέσεων Natura 2000 ε, ε, αποτελούν κυρίως την αρμοδιότητα των ε, ελεγκτικών περιβαλλοντικών ερχών και επομένως θα πρέπει να έχει την εποπτεία η Κομισιόν αλλά θα πρέπει να πιέζει από την άλλη πλευρά και τα κράτη-μέλη έτσι ώστε οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις να είναι καλύτερες. Δεύτερη σειρά ερωτήσεων αφορά το γενικότερο θέμα της χρηματοδότησης και της παρακολούθησης ερώτηση λοιπόν πώς είναι δυνατόν να μειωθούν ε, τα χρηματοδοτικά κενά όσον αφορά την ε, βιοπικιλότητα και πώς θα ενταχθεί η βιοπικιλότητα στον προϋπολογισμό ε, του 2020 γιατί τώρα δίνουμε, παίρνουμε χρήματα και τα παίρνουμε από την ανάπτυξη της υπαίθρου, από τη γεωργία και μετά χρησιμοποιούμε άλλα κονδύλια για να καθαρίσουμε αυτά που έχουν ε, ε, αποκτήσει προβλήματα κατά κάποιο τρόπο λόγω διαφορετικής ε, χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά κονδύλια. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε περισσότερο τα ζητήματα της βιοπικιλότητας και οι πολιτικές μας όπως και τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα να είναι πιο συνοπτικά και λογικά. Επίσης, Βεβαίως ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι την βιοπικιλότητα στο γενικό προϋπολογισμό και το γενικό ε, σχέδιο χρηματοδοτήσεων, αλλά θα πρέπει να ε, υπάρξει και μία χρηματοδότηση η οποία θα αφορά συγκεκριμένα το θέμα αυτό. Ας πούμε λέμε ότι 20% του προϋπολογισμού θα αφορά κλιματικά θέματα. Ε, θα πρέπει να ε, υπάρξει και κάτι αντίστοιχο για την ε, περίπτωση το... της βιοπικιλότητας πέρα από το Life και Life Plus. θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε τα χρήματά μας να χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο και όχι απλώς για να βελτιώνουμε αυτά τα οποία με άλλα κονδύλια ευρωπαϊκά έχουμε καταστρέψει. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Πρόκειται για ένα, μια συζήτηση από την οποία προκύπτουν πολλά ερωτήματα, κυρίως όμως προς την πλευρά της ε, Κομισιόν. Έχουμε τον κύριο Ρικάρδο Λόσα, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που θα μπορούσε ενδεχομένως ε, να απαντήσει στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ, ε, κύριε Πρόεδρε, και ζητώ συγγνώμη που έφτασα με καθυστέρηση. Θα ομαδοποιήσω τα σχόλιά μου και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα απαντήσω στις περισσότερες από τις ερωτήσεις που απήντησα που ε, ε, άκουσα για την Κομισιόν. Πρώτα απ' όλα να πω ότι καλωσορίζει η Κομισιόν αυτήν την ειδική έκθεση γιατί ευθυγραμμίζεται μάλλον με τον έλεγχο κατάστασης fitness check ε, που έκανε η Κομισιόν. Δηλαδή το κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι είναι καλό το πρόγραμμα αλλά χρειάζεται καλύτερη υλοποίηση. Είναι αλήθεια ότι ο τρόπος με τον οποίο υλοποιήθηκε σε πολλές περιπτώσεις ε, το Natura 2000 ε, δεν ε, έδωσε τις πλήρες δυνατότητες στο πρόγραμμα. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιωθούν τα ελαττώματα του παρελθόντος, να μειωθούν τα κενά και επομένως να μπορέσουμε πραγματικά να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που είχαμε μέχρι τώρα αυτό που είδαμε ε, στο κείμενο της 27ης Απριλίου είναι ότι καλύτερη υλοποίηση των οδηγιών ε, θα μας οδηγήσει και σε βελτιωμένη αντίσταση όσον αφορά την βιοπικιλότητα έτσι όπως αυτό ορίζεται στο νέο πρόγραμμα 2014-2020 και με τον τρόπο αυτό θα, θα έχουμε και μια πιο ε, λογική συνολική αντιμετώπιση των προγραμμάτων. Ε, βλέπουμε επίσης ότι αυτή η λογική αντιμετωπίζεται και από το σχέδιο δράσης ε, το οποίο εγκρίθηκε πρόσφατα. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης της Κομισιόν το ε, ε, έχουν, έχει προκύψει από την Κομισιόν, από την εργασία των εμπλεκομένων ε, επιτρόπων και από συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που σχετίζεται με την βιοπικιλότητα έχει ληφθεί σοβαρότατα υπόψη σε αυτό ε, το σχέδιο δράσης όπως επίσης και η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου την οποία συζητούμε τώρα το σχέδιο δράσης θα καλύψει δράσεις ε, που θα υλοποιηθούν ήδη από φέτος ε, μέχρι το 2019. Και να πω και κάτι άλλο, να το ξεκαθαρίσω λοιπόν, το σχέδιο δράσης ε, ούτε θέλει ούτε μπορεί να προδικάσει τις συζητήσεις για το επόμενο πολιετές πλαίσιο ούτε και την μελλοντική συζήτηση για το μέλλον της κοινής γεωργικής πολιτικής. Ξέρετε ότι έχουμε τέσσερις κύριες ε, προτεραιότητες, καλύτερη συνοχή και ε, παροχή οδηγιών. Ε, δεύτερον, το θέμα της οικειοποίησης, ένα σημείο το οποίο θα αφορά την ενδυνάμωση των συνεργειών και τέλος την καλύτερη και αποτελεσματική γενικότερη εμπλοκή. Θα πω δύο λόγια για τα τέσσερα αυτά θέματα. Πρώτον, αυτό που θέλουμε ε, να αφαιρέσουμε από τα κράτη-μέλη ή να τα βοηθήσουμε, να τα προτρέψουμε να αφαιρέσουν είναι ε, το υπερβολικό άχθος έτσι ώστε ε, να υλοποιηθούν οι οδηγίες ε, χωρίς πρόβλημα. Επομένως, στο πρόγραμμα δράσης ε, προβλέπεται η απλούστευση και η ενδυνάμωση των διαδικασιών όσον αφορά την προστασία των ειδών και προβλέπονται επίσης και μηχανισμοί στήριξης για τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να μπορέσουν να εναρμονίσουν τις διαδικασίες τους. Ε, αυτό αφορά και ανταποκρίνεται μάλλον και στις συστάσεις και του εισηγητού ε, και του ελεγκτικού ε, συνεδρίου και θα μεταφραστεί βεβαίως και σε όλες τις γλώσσες. Επίσης, ανταποκρινόμαστε και τις συστάσεις που αφορούν την βελτίωση ε, των ε, ε, αρχών και θα υπάρξουν οπωσδήποτε και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, οδηγίες σε σχέση με το άρθρο 6 της οδηγίας. δεν υπάρχει πουθενά καμία αναφορά που να απαγορεύει την δημιουργία εγκαταστάσεων ε, διαχείρισης ε, και εξυγίανσης των υδάτων. Τρίτον, δημιουργία πράσινων χώρων, ναι, αλλά εδώ ε, ένα κεντρικό στοιχείο του σχεδίου δράσης είναι το εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να βοηθήσουμε και να προτρέψουμε όλες τις, όλα τα ενδιατήματα να έχουν σχέδια διατήρησης και συντήρησης ε, αλλά πάντα με ε, ε, συζήτηση και διαβούλευση με τους εμπλεκομένους και κυρίως δε με τους ιδιοκτήτες της γης. Γιατί πιστεύω ότι αυτή η συνενετική προσέγγιση μόνο καλή μπορεί να είναι για όλους. Επομένως η Κομισιόν θέλει να ενδυναμώσει οπωσδήποτε, αλλά θέλει και συζήτηση και διαβούλευση με τα κράτη-μέλη και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό καλύπτουμε ε, πολλά από τα στοιχεία που αναφέρουν στην ειδική έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου αλλά και τα μελήματα του ε, εισηγητού. Το σχέδιο δράσης επίσης ε, ε, έχει συγκεκριμένες δράσεις για την βελτίωση της γνώσης ε, και την ευκολότερη πρόσβαση στα στοιχεία και τα δεδομένα. Όλα αυτά βρίσκονται στο σχέδιο δράσης και όλα αυτά επιτείνουν τον καλύτερο συντονισμό. Τέλος, το κεντρικό στοιχείο ε, το, είναι το σχέδιο δράσης ε, το οποίο ε, οπωσδήποτε θα προσπαθήσει χωρίς να προδικάζει το πολιετές πρόγραμμα θα προσπαθήσει λέω να φέρει κάποιες καλύτερες συνέργειες ανάμεσα στις διάφορες μορφές χρηματοδότησης. Θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν τις ετήσιες επενδυτικές δομές ε, και θέλουμε καλύτερη υλοποίηση των παύσεων των πλαισίων δράσεων προτεραιότητας, ε, ε, βεβαίως ε, τα σχέδια συντήρησης είναι πάρα πολύ σημαντικά όπως εξάλλου και τα σχέδια διαχείρισης και φυσικά τα κράτη-μέλη είναι αυτά τα οποία μέσω μοιρασμένης διαχείρισης θα μοιράσουν τα κονδύλια αλλά μας ενδιαφέρει να υπάρχει συντονισμός ανάμεσα στα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας, τα ΠΑΦΣ, την χρηματοδότηση και όλα αυτά αυτά τα οποία σχετίζονται ε, με, τους, ε, ε, με τα ενδιατήματα. Επίσης, οι δείκτες, αυτό αναφέρεται σαφέστατα στην ειδική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Το θέμα των δράσεων λοιπόν, συγκεκριμένων δράσεων, την 10 για τα πουλιά, την 11 για, τα, σε, για τους πόρους, σε όλες τις περιπτώσεις παρέχονται νέοι, νέοι δείκτες. Αργότερα, στο, ε, αργότερα μέσα σε αυτή τη χρονιά όμως ε, θα υπάρξουν και εξειδικεύσεις ε, προγραμμάτων καθώς επίσης και κάποιες τροπολογίες, τροποποιήσεις ε, οι οποίες ε, θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη ε, να δημιουργήσουν συνέργειες ανάμεσα στο LIFE και το Natura και στο σχέδιο δράσης μάλιστα φαίνεται και μια μετατόπιση πάνω της τάξης του 10% από το ένα στο άλλο. Ε, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, είναι πάρα πολύ σημαντική, ε, σημαντικό αυτό το σχέδιο δράσης, ενέχει και την εμπλοκή των πολιτών και άλλωστε πλέον ε, η 21η Μαΐου ε, ανακηρύσσεται η μέρα της φύσης και η μέρα του Natura. και ε, με συγκεκριμένες δράσεις υποστηρίζουμε αυτά τα οποία έχουν αναφέρει και το ελεγκτικό συνέδριο αλλά και ο εισηγητής όσον αφορά τη στήριξη που πρέπει να παρασχεθεί στα κράτη-μέλη. Θέλουμε ε, να ενδυναμώσουμε τους ε, δεσμούς μάλιστα ανάμεσα στην βιοπικιλότητα, τη διατήρηση του περιβάλλοντος και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ ε, σημαντικά θέματα και ε, βεβαίως τελειώνοντας να πω ότι θεωρούμε ότι πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να λειτουργήσει καλά το σχέδιο δράσης. Δεν είναι μόνο θέμα της Κομισιόν, ούτε η Κομισιόν από μόνη της μπορεί να υλοποιήσει ε, ε, το σχέδιο αυτό δράσης. Να σας πω ότι θα υπάρξει μία διάσκεψη την 6η Ιουνίου όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα ε, είναι παρόντες ε, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα έχω ένα ερώτημα ανακοινώσατε ότι ε, στις 6 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το, επεξεργασμένο, το ε, επεξεργασμένο action plan. Θα μπορούσαμε να έχουμε και τις κατευθυντήριες ε, για την διαδικασία λήψης αποφάσεων, διότι είναι κάτι το οποίο επήγει ως, καθότι έχουμε ως έτος στόχο το 2019. Όχι, δεν εννοούσα ότι στις 6 Ιουνίου θα είναι έτοιμη οποιοδήποτε καινούργια καθοδιοίκηση. Απλώς ε, παρουσιάζουμε το συνολικό σχέδιο δράσης με όλα του τα τμήματα. Και θα δείτε ότι πολλά θα πρέπει να συζητηθούν γιατί όντως έχουμε διαφορετικές ε, δράσεις. Ε, αλλά άμα τις συνυπολογίσετε όλες πάμε πάνω από, πάνω από τις 100. Όμως σε κάποιε θα κινηθούμε πιο γρήγορα, άλλες θα ε, μας πάρουν περισσότερο χρόνο, αλλά αυτό είναι μία από τις προτεραιότητε να μην ξεχάσουμε την καθοδήγηση, δηλαδή σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Μάλιστα, να δώσουμε το λόγο και πάλι στο Ελεκτρικό Συνέδριο για τα τελικά σχόλια. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα, σε ό,τι φορά ορισμένε παρατηρήσει ε, του Ιρλανδού Ευρωβουλευτή, Ήδη έχουμε απαντήσει. λεπτό δώσουμε. Ε, the ε, the project... Λοιπόν, υπήρχαν ε, έργα και λέμε ότι αν υπάρχει αρνητική αξιολόγηση Αν λοιπόν έχουμε αρνητική αξιολόγηση για ένα μεγάλο έργο, αυτό υπόκειται στις ε, αρχές ε, του γενικού δημοσίου συμφέροντος. Εάν δεν έχουμε εναλλακτική λύση και υιοθετώντα αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό το έργο λοιπόν μπορεί υπό αυτές τις συνθήκες να προχωρήσει. Υπάρχει λοιπόν λύση Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να προχωρήσουν προγράμματα ακόμα και αν έχουν αρνητική αξιολόγηση στο Natura 2000. And... Άλλα σχόλια ή μόνο αυτό θέλατε να πείτε. Βεβαίω θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τις εξαιρετικά χρήσιμες ε, συστάσεις του και όλους εσάς για το μεγάλο ενδιαφέρον ε, που δείξατε για αυτή την έκθεση. Ένα από τα κύρια συμπεράσματα και μηνύματα που αντλούμε από αυτή την έκθεση είναι ότι απαιτείται μια σωστή υλοποίηση ε, του Natura 2000. Και για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει πραγματικό συντονισμό μεταξύ των αρμοδίων αρχών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Και μια ευρεία συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Βέβαια, εξέβρεση καλύτερων συνεργειών μεταξύ ευρωπαϊκών ε, ταμείων και καλύτερη εκτίμηση και λογιστικός έλεγχος ε, των, του κόστους. Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει και πάλι ο εισηγητής για τα καταληκτικά του σχόλια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, συνάδελφοι, γιατί εδώ και καιρό ασχολούμαι με αυτό το ζήτημα και όταν άκουσα ε, τα συγκεκριμένα σας σχόλια διαπίστωσα ότι αυτή η έκθεση ανήκει και σε εσάς, γιατί είστε κι εσείς ε, οι δήμονες σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε λοιπόν ε, εκθέσεις του ελεκτικού συνεδρίου με τις οποίες, τις οποίες εξετάζουμε και καταλήγουμε σε συστάσεις. Αυτή είναι η δουλειά μας. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, τα συμπεράσματα, έχω τρία βασικά συμπεράσματα. Πρώτον, τα κράτη-μέλη δεν ε, συνεργάζονται το ένα με το άλλο και όλοι παρεμβαίνοντας είπαν ότι θα πρέπει να διορθωθεί αυτή η κατάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ε, ίσως έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει. Πρέπει όμως ε, να εξετάσουμε αυτό το ζήτημα. Ιδίω αυτό που είπε ο συνάδελφο, ότι δεν γνωρίζει δεξιά τύπη ή αριστερά. Πρέπει λοιπόν ε, να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση που δεν ξέρει μια χώρα τι κάνει η γείτονα. Εμείς λοιπόν χρηματοδοτούμε ε, προγράμματα που αφορούν ε, διάφορες περιοχές. Ε, μπορούμε να τα συζητούμε, αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Κάποιες φορές έχουμε αντιφατικά στοιχεία και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να διορθωθεί. Μετά, τα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει περισσότερε πρωτοβουλίε. Τα κράτη-μέλη δεν συνεργάζονται μεταξύ του. Η Κομισιόν, λοιπόν, πρέπει να το πούμε ότι πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη για να δουν τι μπορούν να κάνουν μαζί. Μετά, αναφέραμε επίσης την προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις προτεραιότητες για την επόμενη προγραμματική περίοδο μέχρι το 2027 και για την, ε, που είναι η προστασία του περιβάλλοντος για να ε, πετύχουμε τους στόχους ε, της συνθήκης των Παρισίων. Ένα από του βασικού πυλώνε λοιπόν είναι το περιβάλλον. Γι' αυτό θέλουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τα όσα κάνουν τα κράτη-μέλη και τα όσα πρέπει να κάνουν για να πετύχουν τους στόχους της διάσκεψης των Παρισίων. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα συμπέρασμα ε, το οποίο μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Και Συμφωνούμε και με τον εκπρόσωπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον οποίο θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω για την εκπόνηση αυτής της εξαιρετικής έκθεσης. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε το Ελληνικό Συνέδριο και για την έκθεση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ήρθε και απάντησε ερωτήσει ε, των μελών, αλλά και τα μέλη για τις εξαιρετικές ερωτήσει. Τέλο, βεβαίω να ευχαριστήσουμε και τον εισηγητή. Και εδώ φτάνουμε στο τέλο ε, της εξέτασης αυτού του σημείου. Το λόγο έχει και πάλι η πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ ε, που μου ε, δίνετε την ε, Προεδρία. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4. Προετοιμαζόμαστε για την επίσκεψη στην Ουάσιγκτον και θα ήθελα να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι θα παραστούμε στην Παγκόσμια Τράπεζα όχι μόνο για να συναντήσουμε την πρώην Αντιπρόεδρο αλλά να συζητήσουμε και τις σχέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό το λόγο προβλέπεται μια συζήτηση με την Γενική Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού ε, για να τεθούν τα σωστά ερωτήματα και να αναφερθούμε στα, στα ε, ε, σωστά ζητήματα. Ευχαριστώ κυρία Καζάροφ. Ε, και το ερώτημα λοιπόν είναι τι πρέπει οπωσδήποτε να συζητήσουμε κατά τη γνώμη σας στην Washington. Παρακαλώ. Ναι, βοηθάτε η η απάντηση ε, ε, θα είναι ε, να συζητήσουμε με βάση τις μακροχρόνιες συζητήσεις, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα, θα συναντηθείτε τόσο στο Παγκόσμιο τρόπεζο όσο και με τους εταίρους μας στον ΟΗΕ. Το πρώτο θέμα που θα πρέπει να αναφερθεί είναι το πώς θα συζητήσετε, είναι το πώς εργάζονται πάνω στα αποτελέσματα του προϋπολογισμού ε, είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει με την Παγκόσμια Τράπεζα ε, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί ε, και στο μέλλον και με τα Ηνωμένα Έθνη τώρα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητάμε ήδη κατά την συνεδρίαση της Άνοιξης. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε περισσότερα για όλο αυτό. Είναι κάτι σημαντικό το οποίο θα πρέπει να αναφερθεί. Όσον αφορά την Παγκόσμια Τράπεζα, γνωρίζετε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία ε, το, ε, όσον αφορά το ε, σύστημα αποκλεισμού το οποίο έχουμε ενσωματώσει ε, στις χρηματοπιστωτικές μας ρυθμίσεις βασίζεται σε αυτό το οποίο έχει η Παγκόσμια Τράπεζα ο διευθυντής μας κ. Βούλπορκ έχει προσκληθεί τον Σεπτέμβρη αν θυμάμαι καλά για να συζητήσει το θέμα αυτό και νομίζουμε ότι είναι ένα πολύ καλό στοιχείο να υπάρξει το ζήτημα της προστασίας των ομάδων μα, το οποίο επίση θα πρέπει, ε, κατά τη γνώμη μα, να συζητηθεί. Ε, συζητάμε ήδη με την γραμματεία σας ε, παρέχοντας ε, τις διάφορες πληροφορίες τις οποίες έχουμε, τις συμφωνίες με την Παγκόσμια Τράπεζα που ζητήθηκαν στο παρελθόν από τη συγκεκριμένη Επιτροπή και θα σας τα δώσουμε όλα αυτά τις επόμενες μέρες μαζί με όλες τις άλλες πληροφορίες και δεσμεύσεις που έχουμε με τους δύο θεσμού φέτος αλλά και στο παρελθόν στο, όλες ε, δεσμεύσεις για να μπορέσετε να προετοιμάσετε τη συγκεκριμένη αποστολή. Νομίζουμε ότι αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία ήδη εμείς συζητάμε μαζί τους ε, και ε, οι δύο ε, θεσμοί έχουν πολύ καλή σχέση όχι μονάχα με εμά, αλλά και με το ελεγκτικό συνέδριο ε, και ε, πιστεύουμε λοιπόν ότι ε, και για το Κοινοβούλιο είναι καλός θεσμός να αναπτύξει αυτήν την σχέση εμπιστοσύνης και ανταλλαγής απόψεων που έχουμε αναπτύξει και εμείς τα τελευταία χρόνια. Ε, το 1999 ήταν η πρώτη συμφωνία πλαίσιο με τον ΟΗΕ, ε, το 2001 με την Παγκόσμια Τράπεζα ε, και οι δύο συμφωνίες το 2014 και το 2015 επανεξετάστηκαν οπότε υπήρξε η μεγάλη μεταρρύθμιση των χρηματοστηρών πιστοτικών ρυθμίσεων. Ε, σας υποστηρίζουμε λοιπόν ε, σε ό,τι ε, χρειάζεστε και σε ό,τι άλλο θέλετε πέραν των όσων σας έχουμε δώσει για να προετοιμαστείτε για αυτή την αποστολή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ε, φυσικά ε, περιμένουμε ε, σε πληροφορίες σχετικά με το πώς θα είναι η συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, όμως θα θέλαμε και πληροφορίες για το πώς θα είναι η συνεργασία, πώς είναι η συνεργασία με την Κομισιόν. Υπάρχουν κάποια σημεία λοιπόν όπου θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε περισσότερο. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι περισσότερη διαφάνεια ε, δεν, ε, το βρίσκουμε, ε, δεν, δεν διαφωνούμε πάνω σε αυτό με βάση τις πληροφορίες που έχουμε, όμως θα μπορούσατε να πείτε κάποιες πληροφορίες πάνω σε αυτό, να εμβαθύνετε σε όλο αυτό διότι δεν μας έχετε δώσει όλες τις πληροφορίες που θέλουμε όσον αφορά την ε, διαφάνεια και συγκεκριμένα όσον αφορά την Παγκόσμια Τράπεζα ε, νομίζω ότι έχουμε μια πολύ καλή σχέση ε, και ε, συνεχή ανταλλαγή απόψεων ε, έχουμε αναπτύξει ένα νέο εργαλείο διαφάνειας για να μπορέσουμε να μοιραζόμαστε όλες τις προφορίες με τους δωρητές αλλά και με εμά κατευθυνόμαστε προς την ορθή κατεύθυνση διότι μπορούμε να έχουμε την πληροφόρηση για τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουμε έχουμε λοιπόν όσον αφορά την εφαρμογή μπορούμε να έχουμε τις ε, προφορίες και μπορούμε να τις μοιραζόμαστε μαζί σας. Είναι κάτι το οποίο επίσης μπορεί να παρουσιαστεί σε εσά, ε, το οποίο είναι καλό όχι μόνο για την ε, Κομισιόν και την συμμετοχή μας στον προϋπολογισμό, αλλά γενικότερα και για τους άλλους δωρητές. Επίσης, ειλικρινά, δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά τη διαφάνεια. Ναι, ίσως ε, να μην το επικοινωνήσαμε όλο αυτό ε, πολύ καλά ε, μέσα, όμω θα φροντίσουμε να το βελτιώσουμε. όμως ε, δεν μπορώ να πω ότι με αυτούς τους ε, δύο οργανισμούς ε, μπορούν σίγουρα να υπάρξουν βελτιώσεις, ναι μπορούν να, οι πληροφορίες με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν να δίνονται γρηγορότερα, όμως οι σχέσεις που έχουμε μαζί τους και οι προσπάθειες που καταβάλουν για να μας δώσουν πληροφορίες όποτε εμείς τις ζητάμε δεν είναι κάτι το οποίο εμείς ε, ε, ε, θεωρούμε ότι δεν πάει καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Στικόφσκι, ο οποίος ζήτησε το λόγο και χαίρομαι το γεγονό που τρεις εκ των εφτάν που θα συμμετάσχουν βρίσκονται στην αίθουσα σήμερα μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν από μισή ώρα δεν ήξερα αν θα πάω ή όχι. Εν πάση περιπτώσει ε, υπάρχει και μια ολόκληρη διαδικασία για τις ε, θεωρήσεις. Ε, να δούμε αν θα δεν ήξερα αν θα υπάρχει και θέση για δεύτερον από το ΕΛΚ. Εν πάση περιπτώσει πριν από μία ώρα με πληροφόρησαν ότι μπορώ να συμμετάσχω στην αποστολή και χαίρομαι ιδιαίτερος. Χαίρομαι ιδιαίτερος ε, γιατί ε, η αποστολή με την ε, Επιτροπή μας αυτή είναι πάντα κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Ξέρω βέβαια ότι δουλεύουμε πάντα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση ε, σε σχέση με την συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Ε, έχουμε πολλά προγράμματα σε μερικές ε, περιπτώσεις και περιοχές εμείς δεχόμαστε κριτική από πλευρά των μη κυβερνητικών οργανώσεων Δηλαδή ακούμε συχνά ότι ε, στα προγράμματα της Παγκόσμιας Τράπεζας ε, υπάρχει ε, διαφθορά και υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες ιδιαίτερα παρουσιάζουν αυτό το πρόβλημα. Να ρωτήσω υπάρχει καλή συνεργασία όσον αφορά τα θέματα αυτά μεταξύ της Κομισιόν και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Mm, Κοιτάξτε, λέει η Κομισιόν, εμείς έχουμε συζητήσει με την Παγκόσμια Τράπεζα το σύστημα έγκαιρης, έγκαιρου, αποκλεισμού, ε, έγκαιρου ελέγχου και αποκλεισμού εφαρμόζεται στα προγράμματα ε, με την Παγκόσμια Τράπεζα, άρα υπάρχει ένας καλός βαθμός προστασίας. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ταυτοποιήσει κάποιο τομέα όπου στον οποίο να έχουμε διμερείς ε, σχέσεις ε, που να υποφέρουν από τις ε, κατηγορίες που μόλις αναφέρατε. Υπάρχουν βεβαίως και συμφωνίες διμερείς μεταξύ της Όλαφ ε, και της Παγκόσμιας Τράπεζας και εν πάση περιπτώσει εφόσον ε, προκύψουν ε, τέτοιου, τέτοιες υπόνοιες οπωσδήποτε έχουμε τη δυνατότητα και οπωσδήποτε προτιθέμεθα να αντιμετωπίσουμε ε, και να μελετήσουμε σε βάθος ε, τις ε, κατηγορίες αυτές. Αλλά για την ώρα δεν έχουν προκύψει, τουλάχιστον δεν έχουμε λάβει γνώση τέτοιων κατηγοριών για τα κονδύλια τα οποία η Παγκόσμια Τράπεζα διαχειρίζεται εξ ονόματός μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχει ζητήσει το λόγο κάποιο άλλο, οπότε τελειώσαμε με αυτό το σημείο ε, της τη ημερησία διάταξη. Συγγνώμη, ο κύριο Πυρίνσκι. Ευχαριστώ πολύ, ζητώ συγγνώμη που είχα ζητήσει το λόγο, αλλά μάλλον έπρεπε να τον είχα ζητήσει πιο πριν. Εν πάση περιπτώσει, και εγώ έχω την αίσθηση ότι το πρόγραμμα είναι πραγματικά πολύ εντατικό άρα χρήζει καλής προετοιμασίας. Υπάρχει και ένα στοιχείο του προγράμματος, το οποίο μας προβληματίζει λίγο. Αναφέρομαι στην ε, ισορροπία χρόνου ανάμεσα στην Παγκόσμια Τράπεζα, στην οποία δίνουμε, αφιερώνουμε μια ολόκληρη μέρα, και το Γραφείο Λογοδοσίας στη δεύτερη μέρα ε, για το οποίο προβλέπουμε δύο ώρες. Εμείς ε, θα θέλαμε να μάθουμε τους τρόπους με, τον, με τους οποίους ε, η λογοδοσία διασφαλίζεται ο τρόπος ε, με τον οποίο καλύπτεται το θέμα αυτό στην εκτέλεση ε, του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού. Επίσης, ε, θέλουμε να δούμε λίγο πώς αντιμετωπίζει το θέμα των δημόσιων προμηθειών, διαγωνισμών, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Ξέρουμε ε, α, επίσης το θέμα της απάτης, γιατί ξέρουμε ότι ε, από την άλλη πλευρά υπάρχει, ε, υπάρχουν πολλές προχωρημένες περιπτώσεις και είναι πολύ μπροστά όσον αφορά τις απάτες. Γι' αυτό θεωρούσαμε ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Υπάρχει δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και, και να συζητήσουμε τέτοια ζητήματα. Επίσης, την τελευταία μέρα που συνεχίζονται οι επισκέψεις είχαμε την ιδέα ε, να έρθουμε σε επαφή με κάποιους περιβαλλοντικούς οργανισμούς ε, ακριβώς για να συζητήσουμε θέματα ε, διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός κτλ. Έχετε άποψη όσον ε, αφορά το θέμα αυτό. Πιστεύετε ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να το τακτοποιήσουμε, να προβλέψουμε κάτι. Υπάρχει χώρος. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, πιστεύω ε, ότι είναι, ε, σωστό ότι είναι προβληματικό το ότι θα περάσουμε μια ολόκληρη ημέρα με την Παγκοσμία Τράπεζα και μόνο δύο ώρες με το ελεγκτικό συνέδριο της, των Ηνωμένων Πολιτειών. Προσπαθήσαμε την τελευταία μέρα να στριμώξουμε και κάτι με τις ΜΚΟ, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμα με ποιες θα είναι αυτές και γι' αυτό το λόγο καλύτερα όχι. Ε, στο ε, Καπιτόλιο λοιπόν μπορούμε να περάσουμε διαφορετικά ε, το χρόνο μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τα στριμώξουμε όλα αυτά, όμως δεν μπορώ να υποσχοθώ τίποτα. Σε περίπτωση που υπάρξουν προτάσεις σχετικά με το ποιες ΜΚΟ θα είναι, Ευχαριστώ να ακούσω. Ευχαριστώ λοιπόν ε, για το ότι ήρθατε ε, και τώρα περιμένουμε ε, να έρθει ο συνάδελφος Μούρεσαν σχετικά με τον Γενικό Προϋπολογισμό. Ελπίζω ότι ο κύριος Μούρεσαν, ο οποίος έπρεπε να είναι εδώ στις 4.30 θα μπει σιγά σιγά. Δεν θέλω λοιπόν να διακόψω την συνεδρίαση παρόλο που βλέπετε μια μικρή συνεδρίαση, μικρή διακοπή. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. liebe kolleginnen und kollegen der kollege ist eingetroffen ήρθε ο κύριος ε, Μούρισαν, ε, έρχεται και ο ε, συντάκτης νομοθότησης μας, ο κύριος Ζέλλα. Σίγκφριτ, ε, έχεις το λόγο, θα, σας, σου πρότεινα να έρθει να κάτσε δίπλα μου. Ναι, ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερος ε, για το γεγονό ότι έχουμε ε, τον ε, συντάκτη τη γνωμοδότηση για το Γενικό Προπολογισμό της Ένωσης για το 2018. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια καλή συνεργασία με την Επιτροπή προπολογισμού και αυτό επετεύχθη με την κοινή συνεδρία που έχουμε. Σε λίγο θα έρθει και ο δικό μα γνωμοδότη. Αρχικά όμω είναι σημαντικό να ακούσουμε που θα πρέπει να επικεντρωθεί ο προπολογισμό. και επίσης ε, θα θέλαμε ε, να δούμε και μερικά από τα δικά μας ε, ζητήματα τα οποία μας αφορούν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι διατέρες που είμαι εδώ σήμερα το απόγευμα. Κάποιοι βέβαια φοβούνται να καθίσουν κοντά στην κυρία Γκρέσλε. Εγώ όμω δεν ανήκω σε αυτού. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα. Σα ευχαριστώ όλου για την πρόσκληση. Πρώτα και κύρια θα ήθελα να κάνω αυτό ακριβώς που μου ζήτησε η Πρόεδρος. Να σας δώσω μια σύντομη επισκόπηση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων που προτείνω εγώ για τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη χρονιά. Όμως μετά θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις για το πού θεωρείτε ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στον ε, προπολογισμό του 2018. Και θα ήθελα η σημερινή μου επίσκεψη να αποτελέσει και την αρχή της συνεργασίας μας ε, κατά τη διάρκεια τη φετινή χρονιά, γιατί τον Μάρτιο υιοθετήσαμε την έκθεσή μου με τι κατευθύντερες γραμμέ για τον επόμενο προπολογισμό. Τώρα περιμένουμε το προσχέδιο του προπολογισμού, το οποίο θα παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Μαΐου και βέβαια το φθινόπωρο θα έχουμε τι διαπραγματεύσει μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με τη συμμετοχή και τη Κομισιόν βέβαια και είναι σημαντικό για μένα να βρίσκομαι σε στενή επαφή μαζί σα για να γνωρίζω και μετά την δημοσίευση του προσχεδίου προπολογισμού της Κομισιόν να ξέρω ποια θα είναι η δική σας γνώμη. Θεωρώ ότι ο ενωσιακό προπολογισμό για το 2018 πρέπει να έχει δύο βασικές προτεραιότητες. Πρώτον, ανάπτυξη και απασχόληση και δεύτερον, ασφάλεια του πολίτη και προστασία του πολίτη. Εδώ θα πρέπει να δώσουμε έμφαση λοιπόν γιατί αυτό αναμένουν και οι πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέσεις εργασίας και ασφάλεια. Και πώς θεωρούμε εμείς ότι θα τα πετύχουμε όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου. Για να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, χρειαζόμαστε βεβαίως μια ισχυρή οικονομία που θα είναι ανταγωνιστική, αξιόπιστη για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι θέσεις εργασία εκεί δημιουργούνται στον ιδιωτικό τομέα, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όχι στον δημόσιο τομέα. Ε, Χωρί να θέλω να προσβάλλω ή να λυπήσω τους ε, δημοσιου υπαλλήλους. Δεν απευθυνόμαστε όμως εκεί. Γι' αυτό ο σκοπό μου είναι να επενδύσουμε στι υποδομέ, στην καινοτομία, στη στήριξη των μικροπιστών επιχειρήσεων, ιδίω στι ιδιαίτερα καινοτόμε επιχειρήσει, στου επιχειρηματίε και στου νέου επιχειρηματίε, για να αντιμετωπίσουμε και την ανική ανεργία προγράμματα που πρέπει να ενισχυθούν. Ορίζουν 2020 για την έρευνα και καινοτομία, διευκόλυνση συνέδρα στην Ευρώπη για τι υποδομέ, κόσμε για τι μικροψηφίε επιχειρήσει, το έρασμο που δεν είναι μόνο σχέδιο ανταλλαγή ε, φοιτητών. Είναι και ένα πρόγραμμα το οποίο τους επιτρέπει και να μάθουν περισσότερα για την Ευρώπη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ενισχύει και τις πιθανότητέ τους να βρουν μια καλή θέση απασχόλησης στην αγορά εργασία. Γιατί τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το 60% των εργοδοτών στην Ευρώπη θέλουν την διεθνή εμπειρία των νέων εργαζόμενων. Όσο περισσότερη λοιπόν διεθνή εμπειρία έχει αποκομίσει κανείς, τόσο το καλύτερο είναι να βρει μια, μια δουλειά για την απασχόληση των νέων. Η σχετική πρωτοβουλία και όπως βλέπουμε και από την αναθεώρηση του ε, πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου θα έχουμε 1,2 δις ακόμα μέχρι το τέλος του ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ. Η νεανική απασχόληση είναι ισχυρή, μεγάλη, ψηλή στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή την πρωτοβουλία. Όμως εγώ ανήκω σε αυτούς ε, που παίρνουν πολύ στα σοβαρά τι συστάσει και τι εκθέσει του ελληνικού Συνεδρίου και λέω είναι πολύ υψηλή η νεανική, η νεανική ανεργία. Πρέπει να συμβάλλουμε για να πέσει. Όμω δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονό ότι το Ελληνικό Συνέδριο λέει ότι είναι μεικτά τα αποτελέσματα αυτή τη πρωτοβουλία μέχρι τώρα. Γι' αυτό είμαι διατεθειμένο να την επικαιροποιήσω και να τη βελτιώσω αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί το 2013 ψηφίσαμε ένα επταετές πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Βάσει των προτεραιοτήτων που θεωρούσαμε ότι θα πρέπει να ιεραρχηθούν. Από τότε όμως είχαμε και κάποιες απρόσμενες εξελίξεις, τρομοκρατία, έλλειψη ασφάλειας, μεταναστευτική κρίση και προσφυγική κρίση. Επομένω, αξιοποιήσαμε όλους αυτούς τους πόρους που είχαμε για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις κρίσεις. Και βεβαίως αυτό πολύ σωστά το κάναμε, γιατί ήταν επίγουσες οι συνθήκες. Καλά κάναμε λοιπόν. Όμω, επειδή η δημοσιονομική μα πορεία είναι περιορισμένη, πρέπει να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση και του τελευταίου ευρώ. Γι' αυτό λέω ναι στην πρωτοβουλία νεανική απασχόληση, όμω πρέπει να δούμε πώ θα τη βελτιώσουμε. Προπολογισμό με βάση τι επιδόσει. Αν δούμε τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε για κάθε ευρώ που έχουμε δαπανίσει, αυτό πάντα θα πρέπει να το κάνουμε σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Δεύτερη προτεραιότητα, η ασφάλεια. Όπω ξέρετε, ιδίω στους τομείς 3 και 4, οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι. Γι' αυτό και τίθεται το ζήτημα πώς μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας χωρίς να δαπανίσουμε περισσότερα χρήματα. Η ενίσχυση των ενωσιακών οργανισμών που άπτονται των εσωτερικών υποθέσεων, Frontex, EASO, Eurojust είναι, και Europol, είναι αυτοί που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση ε, του ελέγχου των συνόρων, θα βελτιώσουν τη ροή πληροφοριών για τα άτομα που, ε, για τα οποία υπάρχουν υποψίες για την τρομοκρατία, για την ε, ε, εμπορία ανθρώπων ή για τη διακίνηση ε, μεταναστών. Πρέπει λοιπόν να αυξήσουμε τον ε, προπολογισμό για αυτούς τους οργανισμούς και να βελτιώσουν τις ικανότητε τους και δυνατότητές τους. Αρκεί βέβαια αυτό να τεκμηριώνεται. Είμαι ανοιχτό λοιπόν σε αυτό και για την υποπροσκευαστική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπή για την, άμυνα, την έρευνα στον τομέα τη άμυνα. Θεωρώ ότι δεν πρέπει δαπανούμε αυτά τα χρήματα ξεχωριστά σε κάθε κράτος μέλος για να πετύχουμε αντίστοιχα ε, αποτελέσματα. Ας τα δαπανίσουμε πάνω αυτά τα χρήματα μία φορά σε ενωσιακό επίπεδο και να μοιραστούμε μεταξύ μας τα ωφέλη. Τα κράτη-μέλη θεωρώ ότι είναι διατεθειμένα να κάνουν κάτι τέτοιο. Όπως ξέρετε και όπως προείπα, η αναθεώρηση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου συνεχίζεται εμείς διπροντευθήκαμε ένα πακέτο με το Συμβούλιο, το οποίο πρώτα και κύρια δίνει μεγαλύτερη ευελιξία στον προπολογισμό και το Κοινοβούλιο ε, έκανε το δικό του μερίδιο, υιοθετήσαμε την ε, συμφωνία. Το Συμβούλιο όμω δεν το υιοθέτησε την περασμένη εβδομάδα στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο απέτησε να αφαιρεθεί αυτό το σημείο από τη μέσα διάταξη μέχρι τις εκλογές ε, στη Μεγάλη Βρετανία. Και πρέπει εδώ να είμαι πολύ σαφή. Η αναστολή η αναβολή κατά δύο μήνες της ε, υιοθέτηση της αναθεώρησης του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου είναι κάτι το οποίο τελικά εντάξει θα το καταφέρουμε. Θα είναι πολύ δύσκολο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει σχέδιο προπολογισμού χωρίς καμία ευελιξία. Αλλά αν η αναθεώρηση του ΠΔΠ υιοθετηθεί κάποια στιγμή μέχρι τις, διακοπές, ε, τις θερινές διακοπές θα τα καταφέρουμε. Όμως πραγματικά βρίσκεται σε κίνδυνο η αναθεώρηση του ΠΔΠ και αν ε, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ξεμπλοκάρει αυτό το φάκελο, υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος να μην έχουμε προπολογισμό για του χρόνου που να αντιστοιχεί στις ανάγκες ε, του 2018. Και το Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό βέβαια θα πληγεί από την έλλειψη της ε, αναθεώρησης του ΠΔΠ γιατί 1,2 δις παραπάνω θα αφιερωθούν στην πρωτοβουλία για την νεανική απασχόληση, 200 εκατομμύρια για τον ορίζοντα 2020 και άλλα προγράμματα θα πάρουν περισσότερη ε, χρηματοδότηση. Και για τον ορίζοντα 2020, να σα πω ότι το 2015 το ΕΒ ήταν ο μεγαλύτερος δικαιούχο υπό αυτό το πρόγραμμα. Για το 2016 δεν έχουμε ακόμα στοιχεία. Πήραν χρήματα περισσότερα από τη Γερμανία που είναι και το μεγαλύτερο κρατός μέλος και βέβαια το πολύ σωστά γιατί είναι πολύ καλά τα πανεπιστήμια και το καθεξής. Επομένως ε, ορθώς παίρνουν ε, πολλά έργα υπό το Horizon 2020. Όμως, όπως ε, έλεγα και προηγουμένω, όλα αυτά θα επηρεάσουν και τα Βρετανικά Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά του ε, κέντρα. Αυτά από πλευρά μου, Πρόεδρε. Ίσως εν συντομία να σταθώ στα καταπιστεύματα, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, η αντιμετώπιση τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση ήταν ένα εγχείρημα άνευ προηγουμένου. Έπρεπε να δράσουμε γρήγορα και κατεπηγόντω υπό τεράστιε πιέσει. Γνωρίζουμε ότι και εμεί στην Επιτροπή Προπολογισμού δηλώσαμε τη δυσαρέσκειά μα ότι μάθαμε από τον τύπο ότι έπρεπε 500 εκατομμύρια ευρώ να δαπανηθούν ε, για την διευκόλυνση για την Τουρκία και μετά μάθαμε ότι ήταν ένα δις ευρώ χωρίς να υπάρχει καμία διαβούλευση με εμά. Αυτό έγινε υπό ειδικέ ε, περιστάσεις, μεγάλη πίεση κτλ. Οπότε τελικά ε, συμμετείχαμε κι εμείς στην εξέβρεση λύσης, όμως είπαμε ότι δεν πρέπει να ξαναγίνει αυτό στο μέλλον. Από εδώ και πέρα είπαμε ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει στι ε, συναντήσει για τα καταπιστεύματα, να μα ενημερώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστηματικά σε ό,τι αφορά τι εξελίξει για τα ταμεία. Το μόνο που απομένει είναι η ε, ε, δεσμεύση των κρατών μελών. Για το μαντάτα, α πούμε, έχουμε ένα τεράστιο ποσό. Υπό δύσκολε συνθήκε, εμεί τηρήσαμε τι δεσμεύσει μα 117 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τώρα έχουν ταπανίσει τα κράτη-μέλη, που είναι πολύ απογοητευτικό. Πρέπει λοιπόν να τα πάνε καλύτερα τα κράτη-μέλη, γιατί απαιτείται και προβλεψιμότητα. Κλείνοντα. Ορθώς δώσαμε περισσότερα χρήματα στο Ταμείο Μαντάντ, στο ε, στην διευκόλυνση για τους, μετα... για τους πρόσφυγες σε Τουρκία και Βόρεια Αφρική. Να μην ξεχνάμε όμως ότι στις χώρες προέλευσης ή στις χώρες διαμετακόμισης η πολιτική ηγεσία πολύ συχνά είναι τμήμα του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από εκεί. Ε, έλλειψη τροφής, ε, νερού, υποδομών παιδείας, περίθαλψης. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε επιπρόσθετου πόρου που θα κατανεμηθούν σε αυτέ τι χώρε που σωστά του δίνουν περισσότερα χρήματα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε λοιπόν τι βασικέ αιτίε τη μετανάστευση, όμω θα πρέπει να ε, τους, να πείσουμε αυτές τις ηγεσίε να θεσπίσουν μηχανισμούς ε, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης και ότι τελικά αυτοί οι πόροι θα φτάνουν στους τελικούς δικαιούχους και να γνωρίζουμε ότι σε πολλές από αυτές τις χώρες η πολιτική τάξη, η άρχουσα τάξη, είναι μέρος του προβλήματος και όχι μέρος της λύσης. Θα μείνω εδώ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι από πλευρά μου, αυτά είχα να πω. Θα ήθελα τώρα με ενδιαφέρον να ακούσω και τις δικές σας απόψεις και σήμερα, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί μου. Ευχαριστώ πολύ. Ε, για αυτήν την ε, σύντομη ε, παρουσίαση που δίνει μια γενική εικόνα. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα γενικό σχόλιο ότι εμείς με την, ε, ε, με τη δική μας επιτροπή δυσκολευόμαστε διότι ε, όταν έρχεται η απόφαση δεν περιλαμβάνονται τα πρώτα, οι πρώτες κατευθυντήριε οι οποίες έχουν ψηφιστεί. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή Προϋπολογισμού λέει ότι τα πρώτα στοιχεία δεν θα συμπεριληφθούν. Με αυτή τη στάση λοιπόν η Επιτροπή Προϋπολογισμού δίνει δυνατότητες ε, κίνησης και ελευθερίας κίνησης για τον προϋπολογισμό. είναι σημαντικό λοιπόν διότι και το τον προπολογισμό θα πρέπει να επιτύχουμε νέα σημεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Θα πρέπει όλα αυτά να λαμβάνονται υπόψη. Ναι, ε, είμαι ε, μέλος και στις δύο επιτροπές και βλέπω ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία είναι ε, σημαντικά και τα οποία συζητήθηκαν και γι' αυτό το λόγο είναι σημαντικό κάποια στιγμή να υπάρχει ένας γνωμοδότης ο οποίος θα επιτρέψει να συμπεριληφθούν νέες ιδέες, κάτι το οποίο δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Πρώτο σχόλιο. Δεύτερο σχόλιο τώρα, ε, πράγματα τα οποία ε, πριν από την συνθήκη της Λισαβόνας ε, περνούσαμε πολύ εύκολα, δεν μπορούμε να τα περάσουμε τώρα, αφορούν τα αποθέματα, διότι τα αποθέματα χρειάζονται τα τρία πέμπτα σε πλειοψηφία, έτσι λοιπόν είναι σχεδόν αδύνατο να εφαρμοστούν και για αυτό το λόγο η ο γνωμοδότης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα αποθεματικά. Ε, γνωρίζω ότι ε, έχουμε μια συμφωνία όπου δεν απαλλάσσεται από το 2009 το Συμβούλιο. Πώς λοιπόν είναι δυνατό ε, να επιτρέπουμε κάτι τέτοιο ως υπεύθυνοι για τον προϋπολογισμό. Είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι έχουν και τον τελευταίο λόγο για τον προϋπολογισμό είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη να μας. Ε, κάτι ακόμα αφορά την ενσωμάτωση ε, των ειδικών αντιπροσώπων ε, στην εξωτερική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το πολεμήσει ο γνωμοδέτης μέχρι και το τελευταίο σημείο. Δεν είναι, να το, δεν είναι δυνατόν να το επιτρέψουμε ως έχει ε, την πέρσι ε, η εξωτερική υπηρεσία ε, δράσης το ανέλαβε αυτό μόνη της. Η ΑΦΕΤ ήταν υπέρ κάτι τέτοιου. Φροντίσαμε να, υπήρξαν, να υπάρξει υποστήριξη γι' αυτό, όμως ξεπεράστηκαν όλα τα χρονοδιαγράμματα και πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να συμπεριληφθεί. Επίσης υπάρχουν ε, και άλλα ενδιαφέροντα ερωτήματα. Νομίζω ότι πριν από δύο ημέρες ε, αποφάσισε η Κομισιόν ε, για την έκθεση κατά της διαφθοράς το οποίο ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια δέχομαι ότι στη συγκεκριμένη έκθεση ε, δεν ήταν η αγαπημένη μας έκθεση όμως ε, είναι σημαντικό να προωθηθεί όλο αυτό το ερώτημα είναι ε, να υπάρξει μία συμφωνία για να συνεχιστεί αυτή η έκθεση να συνεχίσει να κατατίθεται διότι ήταν, θα ήταν μία δυσάρεστη είδηση εάν κάτι το οποίο ε, ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και το παρουσιάσαμε στο ε, κοινό να πούμε ξαφνικά ότι αδιαφορούμε. Είναι κάτι όμως ε, για το οποίο χρειαζόμαστε την υποστήριξη της Επιτροπής Πλοϋπολογισμού. Πολεμήσαμε από κοινού μία φορά και είχαμε επιτυχία όσον αφορά τις ομάδες ΕΞΠΑΤ και πράγματι ε, καταφέραμε να υπάρξουν αλλαγές. Αν λοιπόν πραγματικά έχουμε μια κοινή γραμμή και οι δύο μπορούμε να εφαρμόσουμε πολλά και να προωθήσουμε πολλά και έχουμε μια ε, μεγαλύτερη δυνατότητα ε, κίνησης. Ε, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά για μένα διότι αν εγκαταλείψουμε τότε δεν θα έχουμε πετύχει τίποτα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σκέφτηκα στα γρήγορα. Στο μεταξύ ήρθε και ο γνωμοδότης ο οποίος θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ε, γνωρίζεις ε, βρισκόμουν σε μια εκδήλωση όπου βρισκόσουν και εσύ πριν από λίγο, οπότε συγγνώμη για όλο αυτό ε, που έρχομαι τώρα. Δεν γνωρίζω τι είπε ο κύριος Μούρεσαν ήδη, όμως από τη δική μας επιτροπή εμείς δεν καταρτίζουμε τον προϋπολογισμό, εμείς εξετάζουμε τι έγινε με τον προϋπολογισμό και την ε, τελευταία εβδομάδα ε, ψηφίσαμε την ε, απαλλαγή όπου αναφέρθηκαν τα ζητήματα για τον προϋπολογισμό του 2015, 15, ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά και για τους επόμενους προϋπολογισμού. Ποια είναι τα βασικά σημεία για το 2014 μέχρι 18. Έχουμε την ε, πέμπτη ε, κατά σειρά ε, χρόνια πώς λοιπόν τα διάφορα προγράμματα εφαρμόζονται πώς γίνεται η στρατηγική, αν ο προϋπολογισμός θέτει τα σωστά κίνητρα αλλά και βάσεις και ταυτόχρονα παρατηρήσαμε ότι έχουμε ε, πώς αντιδράσαμε σε ε, ξαφνικές ε, προκλήσεις όπως είναι, όπου δημιουργήθηκαν για παράδειγμα σχεώδεις προϋπολογισμοί, παράλληλοι προϋπολογισμοί με βάση τη χρηματοπιστωτική κρίση υπήρξε συγχρηματοδότηση για όλο αυτό θέσαμε την στρατηγική και ε, μπορούμε να βρούμε αν ε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις στρατηγικές επενδύσεις ε, θα πρέπει να συμπεριληφθεί σε αυτό. Χρειάζεται μια οικονομική βάση αν ε, θα ε, αφαιρεθεί από τον προϋπολογισμό ή όχι και ποιοι τομείς θα συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Τώρα όσον αφορά ε, τις δόσεις έχουμε καταλήξει στο 18%, το 80% όσον αφορά τις άμεσες επενδύσεις, τις πληρωμές και θα πρέπει να εξετάσουμε που ακόμα ο προϋπολογισμός μπορεί, έχει, διαθέτει ελευθερία κίνησης ε, γνωρίζουμε τις θέσεις του Συμβουλίου όσον αφορά ε, τις ε, δεσμεύσεις για πληρωμές και όσον αφορά τις πιστώσεις που έχουμε όλα αυτά έχουν συζητηθεί στο, στην περίπτωση του προπολογισμού για το 2015 συνειδητοποιήσαμε ότι οι πιστώσει ήταν ε, πολύ μεγάλε και όλα ε, τα κράτη-μέλη και οι συνάδελφοι ζητούν περισσότερα χρήματα όμως ε, τα χρήματα αυτά θα πρέπει να επιστρέφουν στους, σε αυτούς που καταβάλουν το περισσότερο στον προπολογισμό εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού θα πρέπει να ρωτήσουμε το πώς θα διασφαλιστεί ότι ότι θα μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε ε, το έργο μας για τον έλεγχο όσον αφορά την ε, διαφάνεια του ε, προϋπολογισμού. Αυτά είναι ε, τα ερωτήματα για ε, την, αναφο... για την απαλλαγή του 2015 ε, και σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού καθώς βρισκόμαστε στη λήξη αυτής της περίοδου. Ευχαριστώ πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μιλήσει ο κύριος Ουγέλ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι υπεύθυνο για τον τομέα δαπανών. Ακούσα πολύ προσεκτικά και τους δύο εισηγητές και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ιδιαίτερα οι δύο προτεραιότητες που ε, αναφέρθηκαν από τον πρώτο εισηγητή, δηλαδή ανάπτυξη ε, και ε, απασχόληση από τη μία και ασφάλεια από την άλλη, οπωσδήποτε του συμμερίζεται η Κομισιόν και οπωσδήποτε θα δράσει αναλόγως. Επίσης σημειώνουμε ότι ε, και το Συμβούλιο συμμερίζεται τις ίδιες ε, προτεραιότητες, επομένως αυτό ε, είναι πολύ καλός ιονός για την περαιτέρω συνεργασία των δύο οργάνων. Βεβαίως συμμεριζόμαστε τον προβληματισμό του εισηγητού σχετικά με τις καθυστερήσεις όσον αφορά την ενδιάμεση επισκόπηση ε, του πολιετούς πλαισίου. Να πούμε ότι δεν υπήρχε πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο. Βεβαίως και το Κοινοβούλιο έδωσε ε, έγκαιρα την ε, σύμφωνη γνώμη του. Υπολογίζουμε ότι ευελπιστούμε ότι στο εγγύς μέλλον θα προχωρήσει η διαδικασία οπωσδήποτε πάντως όχι πριν από την έγκριση του προσχεδίου προϋπολογισμού από την ε, Κομισιόν. Θα αντικατοπτριστεί η κατάσταση αυτή στον ε, προϋπολογισμό και ενδεχομένως θα πρέπει μετά το καλοκαίρι να έχουμε μια διορθωτική ε, επιστολή έτσι ώστε να ενταχθεί και το θέμα αυτό. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι άλλο να πω για την ώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ ε, πολύ. Κατά από ό,τι φαίνεται όλοι ε, ε, λείπουν σήμερα. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Σίγκβαιτ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα κυρία Πρόεδρε. Είναι γι' αυτό ακριβώς εγώ έρχομαι σε επαφή και επισκέπτομαι όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές έτσι ώστε να ανταλλάξω απόψεις, να συλλέξω ιδέες κλπ. Κυρία Πρόεδρε, πραγματικά τώρα είμαι σε φάση ε, ε, που προσπαθώ να συλλέξω στοιχεία, να ακούσω προσεκτικά, ε, ακούω προσεκτικά και τον εισηγητή σας θα πρέπει προς το τέλος ε, του χρόνου να κάνουμε ε, την ε, τελική αξιολόγηση, να δούμε δηλαδή αν έχω καταφέρει τελικά κάτι. Αλλά Όσον αφορά τους εξωτερικούς ε, ε, συμβούλους της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί, θα πρέπει να το δούμε. Τα καλά νέα είναι ότι ε, για φέτος τουλάχιστον προλαβαίνουμε τις προθεσμίες, το έχω συζητήσει και με τους συναδέλφους της ΑΦΕΤ. Δεύτερον, σε σχέση με τα όσα είπε ο εισηγητής όσον αφορά το ποσοστό απορρόφησης και τα σχετικά στοιχεία. Αλήθεια είναι ότι το ποσοστό απορρόφησης στα περισσότερα κράτη-μέλη είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δεν ξεκολλάει, δεν απογειώνεται η ε, διαδικασία και φαντάζομαι ότι το 17 θα είναι παρόμοιο με το 16, δηλαδή ότι όλα τα ποσά τα οποία ε, ε, βρίσκονται εκεί προς απορρόφηση δεν θα ε, απορροφηθούν όλα, θα παραμείνουν αποθεματικά και βεβαίως ξέρουμε ότι σε ορισμένες περιφέρειες και σε ορισμένα κράτη-μέλη ε, θα υπάρχουν προβλήματα ε, όσον αφορά τις ε, πληρωμές ήδη από τις 564 ρυθμιστικές αρχές μονάχα 351 έχουν πιστοποιηθεί δηλαδή έχουμε περίπου 100 και πλέον αρχές οι οποίες δεν έχουν πιστοποιηθεί υπάρχουν όμως και χώρες όπως ας πούμε στην Ρουμανία όπου μονάχα δύο από τους 10 οργανισμούς έχουν, έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αυτό είναι πολύ κακό, ενώ υπάρχουν και άλλες χώρες όπου το ποσοστό είναι ε, αντίστροφο. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε πώς έχει η κατάσταση ε, όσον αφορά τις πιστώσεις πληρωμών, γιατί είδαμε ότι τα προγράμματα δεν προχώρησαν αρκετά το 2016 και επομένως οι πιστώσεις υποχρεώσεων ήταν πολύ ψηλότερες από τις πιστώσεις πληρωμών. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τις υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από τις συνθήκες και θα πρέπει να ε, ε, ε, αποφασίσουν να συμβάλλουν, συγγνώμη, να συνενέσουν οι χώρες έτσι ώστε να ξαναμπούν τα χρήματα αυτά στο προϋπολογισμό. από την άλλη πλευρά, εάν μας ζητηθεί να κάνουμε κάτι περισσότερο με τον ίδιο προϋπολογισμό μπορεί ενδεχομένως να εντείνουμε τις προσπάθειες εντός των, ε, ε, προσδιάθεση, των διαθεσίμων κονδύλιων, αλλά ε, το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιες προτεραιότητες, τις οποίες δεν είχαμε προβλέψει το 2013. Σίγουρα υπάρχουν θέματα όπως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είναι η γεωργία που τις ξέραμε, είναι παλιές προτεραιότητες, αλλά προκύπτουν και νέες προτεραιότητες, οι οποίες χρειάζονται και αυτές χρήματα ε, για να ολοκληρώσω όσον αφορά ε, τα επενδυτικά ε, ταμεία και τα ταμεία ε, συνοχής, ξέρετε ότι η ε, ε, πήραμε χρήματα και από τον ορίζοντα 2020 ε, και από την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει και συζήτηση στην Κομισιόν για τον ορίζοντα 2020 πολλά από τα προγράμματα τα οποία έχουν ε, χρηματοδοτηθεί από το ΕΦΣΥ ε, κατά 35% σύμφωνα με την Κομισιόν και τον Αρμόδιο Επίτροπο 35% ε, των προγραμμάτων έχουν ένα σκέλος προχωρημένης τεχνολογίας Επίσης 500 εκατομμύρια, ε, εάν συνεχιστεί ο προγραμματισμός ως έχει, ε, θα ε, ληφθούν από την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Ο συνάδελφος ε, Ούντο Μπούλμαν ε, έχει ε, καταλήξει στο συμπέρασμα στην έκθεσή του ότι δεν έχει, υπάρχει, δεν έχει υπάρξει για την ώρα πρόβλημα όσον αφορά την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη μετά από την έγκριση του ΕΦΣΥ. Αλλά βλέπουμε ότι στα δύο πρώτα χρόνια αυτού του πολυετούς προγράμματος η απορρόφηση είναι 13% σε σχέση με το 19% που είχαμε ε, στο προηγούμενο πολιετές ε, πλαίσιο. Επίσης είναι σαφές ε, λόγω του, της δημιουργίας του ΕΦΣΙ έχει προβλήματα και το πρόγραμμα Horizon 2020 δεν έχουν ενταχθεί εκεί όλα τα προγράμματα που θα θέλαμε δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτά που στο παρελθόν έχουν χρηματοδοτηθεί γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό αυτό που στο πολιετές ε, πλαίσιο προσθέτει 200 εκατομμύρια ε, στο ε, ορίζοντα 2020. και θα δούμε κατά πόσον μετά από την προσθήκη των νέων κονδυλίων θα έχουμε κάποιο περιθώριο κάποιο περιθώριο ευχέρειας ε, θα δούμε πώς θα έχουν τα πράγματα και βεβαίως πιο συγκεκριμένα θα μιλήσουμε όταν έχουμε το προσχέδιο από πλευράς της Κομισιόν. Μην φοβάσαι, Σίγκριτ, δεν έχω ερωτήσει. Είμαι ο μοναδικό ευρωβουλευτή εδώ πέραν ε, τη Προέδρου και του εισηγητή. Α, ναι, και εσεί. Τέλο πάντων, δεν είμαστε πολλοί. Όμω, ήθελα απλώ να σα ενθαρρύνω λιγάκι. Βεβαίω, ε, απασχόληση και ασφάλεια. Δεν θέλω να επιστρέψω στι λεπτομέρειε γιατί εδώ έχουμε τα ζητήματα του προπολογισμού. Να πω όμω το εξή. Όταν είπατε ότι αυτό θέλουν οι πολίτε. Το είπατε προηγουμένω. Εγώ λοιπόν σα ενθαρρύνω πραγματικά να προσπαθήσετε και να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας Ξέρω βέβαια ότι ήδη έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες και ότι υπάρχουν και συγκεκριμένες ε, συγκυρίες και συνθήκες. Αλλά να κάνετε ό,τι μπορείτε για να γίνει αυτό το πράγμα όσο το δυνατόν πιο αντιληπτό από τους ε, πολίτες. Το 2018 λοιπόν θα είναι ένα έτος, θα έχουμε έναν προπολογισμό το οποίο θα πρέπει πραγματικά να έχει πρακτικές ε, προεκτάσεις για τους πολίτες. Για το θέμα των δημοσιονομικών περιορισμών με βάση και τα όσα είπε η Πρόεδρος, κυρία Γκρέσλε. Ο δημοσιονομικός έλεγχος δεν άπτεται μόνο της νομικής ε, πτυχής και όλο ένα και περισσότερο, και εδώ είναι και η αλληλεπικάλυψη ε, μεταξύ της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Προπολογισμών. Ε, λοιπόν, αλληλεπικάλυψη λοιπόν μεταξύ επιδόσεων και αποτελεσμάτων. Στο ίδιο καζάνι βράζουμε λοιπόν, γι' αυτό και σας ενθαρρύνουμε και ελπίζω τώρα που έχουμε και τον νέο συγητή εδώ για τον προπολογισμό να έχουμε όσο το γίνεται μεγαλύτερη συνεργασία μαζί με την ευελιξία για να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε με βάση τον προπολογισμό που αναφέρατε. Και πιστεύω ότι εδώ μπορούμε να τα πάμε καλύτερα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ευχαριστώ. We Συμφωνούμε απολύτω. Κύριε Τσάιλερ, θέλετε να πάρετε το λόγο. Εκτός μικροφώνου μιλητής. Yeah. Jetzt ist an. Τώρα μάλιστα. Ε, λοιπόν, ε, ακόμα ε, βρισκόμαστε στη διαδικασία των συζητήσεων. Ευχαριστούμε που παρευρέθηκε εδώ πέρα ο κύριος Μουρεσάν. Ναι, ε, η Επιτροπή του θα πρέπει να, να δώσει τις κατευθυντήριες και στη συνέχεια εμείς ε, με βάση αυτές τις κατευθυντήριες ε, όπως είπε και ο Πέτρη θα πρέπει να φέρουμε αποτελέσματα και για να είναι αυτό αρκετά σωστά συνεργαζόμαστε και σίγουρα θα έχουμε και άλλες δυνατότητες ανταλλαγής απόψεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και έτσι λοιπόν φτάσαμε και στο τέρμα αυτού του σημείου της ημερήσιας διάταξης και ευχαριστώ πολύ και περνάμε τώρα στο ε, σημείο 7 το οποίο αφορά την ε, Μολδαβία. Ε, στις 15 ε, Απριλίου διαβάσαμε μία συνέντευξη του Προέδρου Ίγκον Ντόλτον, ο οποίος δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2007 με το 2015 έχει υποστηρίξει με 782 εκατομμύρια την Ευρωπαϊκή Ένωση, την στην Μολδαβία το οποίο ισχύει, το ελέγξαμε όμως ε, πάνω από το μισό αυτό των ε, χρημάτων έχει ε, χαθεί σε σκοτεινά μονοπάτια ε, είναι λοιπόν μια ασυνήθιστη στάση ο, ε, ε, ο πρόεδρος μιας χώρας να ισχυρίζεται κάτι τέτοιο το διαβάσαμε στην εφημερίδα και είναι αναγκαίο λοιπόν να συζητήσουμε και όλο αυτό σήμερα επίσης είπε ότι οι πληρωμές από τη Δύση θα μπορούσαν να ήταν πιο στενά συνδεδεμένες με προϋποθέσεις και να υπάρχουν διμερείς δάνεια και υπάρχουν διμερεί δάνεια τα οποία έχουν πέσει σε λάθος ε, χέρια. Ε, όταν ακούμε για διμερή δάνεια ε, τότε σκεφτόμαστε το δούνου του το οποίο έχει δώσει 15 εκατομμύρια δολάρια στην Μολδαβία το οποίο είναι ένα αρκετά πασό και το ερώτημα λοιπόν είναι τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδώ πέρα και πώς ε, θα το αξιολογήσουμε όλο αυτό. Ε, υπήρξε έκθεση από την ε, πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου, ωστόσο δεν μπορέσαμε να διαβάσουμε όλα τα σημεία. Θέλουμε λοιπόν να λάβουμε και άλλες πληροφορίες από την Γενική Διεύθυνση Γειτονίας και ε, από την Γενική Διεύθυνση ε, Γειτονίας ε, έχουμε 12 εκατομμύρια από το ίνι 70 εκατομμύρια διότι μιλάμε για 36 εκατομμύρια τα οποία έχουν χαθεί. Ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, οι παρατηρήσεις ε, του Προέδρου Ντοντών ε, προσέλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών. Αναφέρατε και εσείς στη συνάντησή του με τη Διβέλτ. Όμως, Τα όσα θα σας ε, αναφέρω τώρα έχουν κοινοποιηθεί και στον κύριο Ντόντον από τον επικεφαλής της αποστολής μας στη Μολδαβία πριν από δύο εβδομάδες. Ακριβώ μετά λοιπόν από τη δημοσιοποίηση τη συνέντευξη, καθώ και στην αρχή τη χρονιά στι Βρυξέλλε, όταν είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο ε, ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την είπατε εκπρόσωπο κ. Μαγκερίνη και τον ε, Επίτροπο Χάν. Πρώτον, μια γενική παρατήρηση για το πώ χειριζόμαστε τι καταστάσει όπω αυτέ με τη Βολδαβία. Όλες αυτές οι εκταμιεύσεις γίνονται μόνο όταν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και συγκεκριμένες συνθήκες που απαιτούν μεταρρυθμίσεις και πρόοδο σε συγκεκριμένου τομεί. Επομένω, ε, καταβάλλονται αυτέ οι εκτεμιεύσει εκ των υστέρων, αναμεταρρύθμιση και εφόσον έχουν υλοποιηθεί μεταρρυθμίσει. Ξέρετε ότι στο παρελθόν έχουμε αποφασίσει ε, να ε, αναστείλουμε για παράδειγμα ορισμένε τέτοιε προσπάθειε στη Μολδαβία. Επομένω, υπάρχουν πολύ ξεκάθαρα κριτήρια τα οποία παληθεύονται κιόλας από εξωτερικού ε, εμπειρογνώμονε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση στι αποστολέ. Σε ό,τι αφορά τώρα τι ε, καταγγελίε του Προέδρου, πρώτον, τα στοιχεία δεν είναι ακριβή. Το ποσό που αναφέρεται, 782 εκατομμύρια, είναι το ποσό το οποίο κατανέμεται στη Μολδαβία για την περίοδο 2007-2015, όπως αναφέρεται εξάλλου και στην έκθεση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Περίπου 87 εκατομμύρια ε, κάθε χρόνο. Και όταν κατανέμεται το κονδύλι αυτό, μεταφράζεται σε δημοσιονομική δέσμευση και βάσει των αποτελεσμάτων κάνουμε τις πληρωμές. Από τα 782 εκατομμύρια λοιπόν, περίπου 63% δίνεται για την ε, ε, στήριξη του προπολογισμού. Αυτό σημαίνει... Τέλος πάντων, έχω πολύ συγκεκριμένα ε, αριθμητικά στοιχεία. Για να μην σας μπερδέψω, μπορώ να σας στείλω και γραπτός. Το 37% λοιπόν πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα, παρόχους υπηρεσιών, μη κυβερνητικέ οργανώσει και διεθνείς οργανισμούς. Όταν λοιπόν το ελεγκτικό συνέδριο ε, εκπώνησε την έκθεσή του, εκείνη τη στιγμή λοιπόν εμείς είχαμε πληρώσει 363 εκατομμύρια, τα οποία σήμερα έχουν φτάσει στα 454 εκατομμύρια, εκ των οποίων 279 είχαν ε, ε, δαπανηθεί για την στήριξη του προπολογισμού. Δεν υπάρχει καμία σύνδεση μεταξύ της απάτης του ενό δις δολαρίων σε τρεις ε, μολδαβικές τράπεζες δεν έχει καμία σχέση με ε, ε, τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Δεν ήταν λοιπόν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, βεβαίως τα έχουμε συζητήσει επί μακρόν αυτά για την κατάσταση στον τραπεζικό κλάδο στη Μολδαβία. και στην συνεδρίασή σας ε, το Δεκέμβρη, ε, το Ελληνικό Συνέδριο συμφώνησε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Μολδαβική κυβέρνηση θα πρέπει να διεξαγάγει τι απαραίτητες έρευνε. Τέλο, αλλά μάλλον αυτό είναι και το πιο σημαντικό στοιχείο, επειδή ήταν μια δημόσια καταγγελία ε, και ο Ευρωπαϊκός Εκπρόσωπος ζήτησε να ενημερωθούν και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα εάν έχει ο Πρόεδρος στοιχεία που να αποδεικνύουν ε, ε, κάποια ε, τέτοια κατάχρηση και εμείς σε αυτή την περίπτωση θα προχωρούσαμε σε, στην υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν για αναστολή των πληρωμών. Όμως δεν μας έχει υποβάλει τέτοια, και προσκομίσει τέτοια στοιχεία ο Πρόεδρος και επειδή το μήνυμά του ήταν τόσο δυσάρεστο και διαβιβάσαμε και εμείς τον Όλαφ όλα όσα γνωρίζαμε για αυτές τις καταγγελίες. όλα Όλαφ διεξήγαγε μια προκαταρκτική έρευνα και κατέληξε το συμπέρασμα ότι το περιεχόμενο του άρθρου δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή αρκετά ακριβές και συγκεκριμένο για να ε, τεκμηριώνεται έτσι η έναρξη μιας ε, έρευνας. Αν όμως λάβουμε οποιαδήποτε νέα στοιχεία που να υποστηρίζουν ε, ε, και να ενισχύουν αυτές τις υποψίες, ε, τότε εμείς βεβαίω θα τα μεταφέρουμε στον Όλαφ. Για το μέλλον τώρα, να ξεκαθαρίσω ότι οι δικές μας υπηρεσίες δεν έχουν προγραμματίσει οποιαδήποτε τέτοια συνδρομή στον ετήσιο πραγματισμό 2016-2017 Εμείς λοιπόν αυτή τη στιγμή εκταμιεύουμε δεσμεύσεις του παρελθόντος, ακολουθώντας και την συμφωνία μεταξύ της Μολδαβικής Κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που συνήθει τον περασμένο Νοέμβριο. Για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο του 2016-2017, εμείς επικεντρώνουμε σε ε, κεντρωνόμαστε μάλλον σε προγράμματα που θα έχουν αποτελέσματα σε τομείς όπως ε, ε, η παροχή υδάτων, απορρίμματα και το καθεξής. Και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και επενδύσεις σε, έναν, σε μια υποδομή διασύνδεσης μεταξύ Μολδαβίας και Ρουμανίας. Με τα χαρά σας θα δώσω όλα αυτά και γραπτός, αν δεν είναι επαρκώς ξεκάθαρα, αλλά είμαι και στην διάθεσή σα για τυχόν περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες, όμως αυτό είναι ε, σάτυρα. Όταν ο ε, αρχηγός κράτους λέει, κοιτάξτε να δείτε, σας εξαπατούμε. Ε, σας ξαπατούμε ε, όσον αφορά τα μισά ε, ποσά που μας δίνετε και στη συνέχεια ζητάμε να γίνετε πιο συγκεκριμένους και στη συνέχεια λέει όχι. Ναι, πρέπει να υπάρχουν συνέπειες για όλο αυτό. Προσβάλλει την ίδια του τη χώρα. Τι συζήτηση γίνεται στη Μολδαβία για όλο αυτό. Δεν είναι δυνατό να έχουμε μια τέτοια δήλωση και να λέμε εντάξει μωρέ αστευότανε». Ε, και δεν ε, είδε τη συγκεκριμένη δήλωση. Το ερώτημα μου είναι αν έκανε κάτι τέτοιο. Ε, ο κύριος Τσέλα έχει κάτι να δηλώσει. Σίγουρα θα πρέπει να εξετάσουμε και το πολιτικό υπόβαθρο όπου το ένα κόμμα προσπαθεί να σκάψει τον τάφο του άλλου το, βλέπουμε ότι στο κοινοβούλιο έχουμε τα, ε, τα κόμματα τα οποία είναι ε, προρωσικά και αυτά τα οποία είναι προευρωπαϊκά ε, και με τέτοιες λοιπόν κατηγορίες προσπαθούν να επιτύχουν κάτι παρόλα αυτά όμως τα όσα έχει πει ο πρόεδρος σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να δώσει και τις αποδείξεις για όλο αυτό διότι ε, αλλιώς ε, είναι κάτι το οποίο γνωρίζουμε από τέτοιες ε, χώρες όπου προσπαθούν με κατηγορίες να υποσκάψουν τον πολιτικό τους αντίπαλο όμως ε, δεν λέμε ότι η Μολδαβία ε, δεν ε, αντιμετωπίζει προβλήματα διαφθοράς. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Πρόσφατα σε μία συνάντηση που είχα με μία συνάντηση σε πανεπιστήμιο όταν πληρώσεις ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να συζητήσεις μαζί του τότε καταλαβαίνουμε ότι ναι, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το πρόβλημα όμως σε αυτές τις ε, βοήθειες είναι ότι δίνουμε το, τα ποστά ε, στον προϋπολογισμό και στη συνέχεια επαφίεται στο ίδιο το ε, κράτος να εξετάζει την εφαρμογή και να κατευθύνει πού πηγαίνουν αυτοί οι πόροι και εμείς θα πρέπει να μάθουμε πού χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα χρήματα και πώς και να έχουμε, να, να έχουμε τη διαβεβαίωση ότι τηρούνται οι κανονισμοί. Ε, το έχουμε βιώσει αυτό και στη Βολιβία με προγράμματα ε, για το νερό που υπήρξε ε, βοήθεια για την ενίσχυση της γεωργίας και όπου η όλη δουλειά έγινε πάρα πολύ καλή όμως η κατάσταση είναι ότι η κατηγορία είναι ότι μονάχα συγκεκριμένες περιοχές και χωριά βοηθήθηκαν ενώ άλλες περιοχές έπρεπε να περιμένουν πάρα πολύ μέχρι να λάβουν βοήθεια και μιλάμε για τα χωριά τα οποία υποστηρίζουν τον πρόεδρο και χωριά τα οποία όμως είναι κατά του Προέδρου. Ε, είναι λοιπόν υποχρέωσή μας να εξετάσουμε ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις ε, με τα μέσα τα οποία ε, διατίθουμε. Η κυρία Κάους τώρα ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ήρθα εδώ πέρα διότι θεωρώ πάρα πολύ καλό το ότι συμπεριλάβατε στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα της Μολδαβίας και με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως το συγκεκριμένο θέμα. Ε, σύντομα ε, στο Κισινάου θα έχουμε την ε, συνεδρίασή μας και σίγουρα θα επανεξετάσουμε το θέμα αυτό. Ε, θα γίνει τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Πιστεύω λοιπόν ότι όπως είπε και ο συνάδελφος μόλις τώρα, όταν ο πρόεδρος μιας χώρας, όπως και αν το αξιολογούμε πολιτικά αυτό το κράτος, δηλώνει κάτι τέτοιο, τότε ε, φυσικά και θα πρέπει να το εξετάσουμε ε, σε σημείο που ε, ακόμα και, στην, ε, και στους πολίτες της χώρας να μπορούμε να πούμε ότι ναι το εξετάσαμε και ξεκαθαρίστηκε ή ότι αυτά είναι τα προβλήματα και έτσι έχει η κατάσταση. Γνωρίζω ότι στην Μολδαβία η διάθεση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει αρκετά ε, σκεπτική διότι η διαφθορά στη χώρα δεν έχει περιοριστεί ε, και αυτό είναι ιδιαίτερα ε, δυσάρεστο λαμβάνοντας υπόψη αυτή τη μεγάλη κλοπή και ε, ταυτόχρονα θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ε, Κομισιόν ε, όταν λέμε όταν κλάπησαν ένα δισεκατομμύρια ένα δισεκατομμύριο αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο ευθυνόμαστε εμείς εμείς θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε ούτω ώστε να ξεκαθαριστεί όλο αυτό διότι είναι ένας μεγάλος σκάνδαλο το οποίο δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ε, και θα πρέπει ε, να ε, πούμε και στον Τόντον ότι και αυτός φέρει ευθύνη ο οποίος θα πρέπει να προωθήσει να υπάρξει μια ξεκαθάριση πάνω πάνω σε αυτό το θέμα Όμω, όλες οι κατηγορίες αυτές που αναφέρθηκαν θεωρώ ότι πρέπει να τις συζητήσουμε επιθετικά ε, και ε, θα πρέπει να εξεταστεί όλο αυτό. Ε, τώρα ποια είναι τα εργαλεία τα οποία έχετε εσείς κυρία Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι. Όμως με ενδιαφέρει ιδιαιτέρω η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την ανατολική γειτονία να μην την αντιμετωπίζουν ως έναν οργανισμό ο οποίος κατηγορίες ε, όσον αφορά την ε, διαφθορά και την αυξαφάνιση δημοσίων πόρων ότι εμείς ε, απλά τέτοιες κατηγορίες τις αγνοούμε. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε το κατάλαβα εν μέρη, όμως δεν θεωρώ ότι είναι καλό και πιστεύω λοιπόν ότι πριν μεταβούμε εκεί πέρα θα πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος συνάδελφος Ιβαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα Το πολιτικό πλαίσιο στην Μολδαβία είναι περίπλοκο. Και μάλιστα είναι περίπλοκο εδώ και αρκετό καιρό. Δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, υπάρχουν κάποιες ε, ε συμμαχίες οι οποίες εμφανίζονται, εξαφανίζονται, δημιουργούνται, διαλύονται. Η κατάσταση λοιπόν είναι από μόνη της περίπλοκη και βεβαίως ε, οι δηλώσεις ε, του νέου Προέδρου ε, της ε, Μολδοβίας ε, Ντοντόνα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στα πλαίσια της εσωτερικής διαμάχης της Μολδαβίας. Βεβαίως τα λόγια του ήταν βαριά και επομένως θα πρέπει οπωσδήποτε να τα λάβουμε υπόψη μας και να κάνουμε τις σχετικές ερευνητικές διαδικασίες. Οπότε άλλωστε το κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε οποτεδήποτε ε, γίνεται λόγος για διαφθορά και οποτεδήποτε χρησιμοποιούνται ε, κονδύλια ευρωπαϊκά και η Επιτροπή μας και η Κομισιόν ε, οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος τα πράγματα. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες που έχουμε ε, ε, βάση των οργάνων συνεργασίας με την ε, Δημοκρατία της Μολδαβίας και όλες οι δικές μου πηγές δεν επιβεβαιώνουν τα λεγόμενα του Πρόεδρου Ντοντών. Ο οικονομικός έλεγχος του ελεγκτικού, Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου επίσης δεν κατέδειξε ε, τη, τους ισχυρισμούς αυτούς. Άλλωστε είναι υποχρεωμένος ο πρόεδρος Δοντών ε, αυτός να παράσχει πληροφορίες ε, σε σχέση με τις κατηγορίες ε, που εξτόμησε. Εμείς πάντα βεβαίως όταν ακούμε τέτοιες αιτιάσεις πρέπει να είμαστε προσεκτικοί γιατί δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία των λόγων του Ντοντών. Ευχαριστώ ο ε, συνάδελφος ε, Σάρβαμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι παράλογο. Τι να σας πω, είναι παράλογο. Ποιο είναι το πρόβλημά μας. Το πρόβλημα είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο έχουμε τέτοια προγράμματα αλλά δεν αρκεί από ό,τι φαίνεται. Στόχο των προγραμμάτων είναι ακριβώ να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να γίνουν σταθερές δημοκρατίες ε, πρώτων συνόρων μας. Γι' αυτό προσπαθούμε να τι βοηθήσουμε. Κατανοώ βεβαίως την πολιτική κατάσταση που ισχύει σε πολλές ε, τέτοιου είδους χώρες. Ωστόσο, έστω και γνωρίζοντας όλα τα στοιχεία αυτά. Το ερώτημα το πραγματικό παραμένει. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Πραγματικά το εννοώ. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Γιατί μας το ζητούν και οι ε, πολίτες μας και οι ψηφοφόροι μας. Αυτοί από τους οποίους έρχονται τα χρήματα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό ερώτημα. Ερώτημα το οποίο εμείς εδώ ως βουλευτές πρέπει να απαντήσουμε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν, με ποιους τρόπους μπορούμε να ενεργήσουμε, έτσι ώστε και σε τούτη την περίπτωση να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Ποια είναι τα απτά μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Φοβούμαι ότι δεν έχουμε και πολλά. Και επομένως το τελικό ερώτημα παραμένει και παρακαλώ ε, να καταβληθούν πραγματικά όλες οι προσπάθειες, να δούμε το, το θέμα από όλες τις δυνατές γωνίες. Εάν δεν έχουμε μέσα στη διάθεσή μας, θα πρέπει να σταματήσουμε και να σκεφτούμε. Αυτό δεν θα το κάνουμε βέβαια σήμερα και σε τούτη τη συζήτηση εδώ. Όλα είναι πιθανά και θα πρέπει να αλλάξουμε τους όρους, θα πρέπει να αλλάξουμε τους κανόνες εάν χρειάζεται να αλλάξουμε ακόμα και την νομοθεσία. Δεν είναι δυνατόν να ε, βρισκόμαστε κατά διαστήματα σε τέτοιες καταστάσεις οι οποίες είναι απολύτως παράλογες και ε, ε, όπου εμείς, εμείς που πληρώνουμε, εμείς που παρέχουμε τα χρήματα να μην έχουμε καμία δυνατότητα να ελέγξουμε. Ναι, αλλά εάν δεν ξέρουμε τι συμβαίνει στη Μολδαβία και αν δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στη Μολδαβία, κάτι θα πρέπει να αλλάξει και κάπως θα πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ναι, σωστά. Πιστεύω και εγώ ότι ε, ε ο πρόεδρος ε, κάνει ένα πολιτικό παιχνίδι αυτή τη στιγμή, όμως εμείς δεν πρέπει να ε, μείνουμε άπραγοι. Ποιο είναι το σχέδιο, πώς θα συνεχίσουμε. δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τα όσα έχουν παρουσιαστεί, όμως πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αρχικά όσον αφορά το πλαίσιο, κύριε Τσέρερ, νομίζω ότι ε, απάντησα το πρώτο σας ερωτήμα ε, η δήλωση του Προέδρου έχει να κάνει με την πολιτική κατάσταση στην ε, Μολδαβία. Έχουμε να κάνουμε μια συγκατοίκηση μεταξύ ενός Προέδρου ο οποίος είναι σκεπτικιστής και από την άλλη έχουμε μια προευρωπαϊκή κυβέρνηση. Βλέπουμε δηλαδή που υπάρχει το πρόβλημα. Ε, και αυτό ήταν ε, και ο λόγος, έτσι το βλέπουμε εμείς. Ο ε, πρόεδρος δεν έδωσε καθόλου αποδείξεις, του ζητήσαμε ε, τόσο διμερός ε, μέσω της διπλωματικής ε, οδού της πρεσβείας μας στο Κισινάου πριν από δύο εβδομάδες αν θυμάμαι ορθά αλλά και στη συνέχεια δημοσίως μέσω της εκπροσώπου της Κομισιόν τον παρακαλέσαμε να μας δώσει αποδείξεις κάτι το οποίο δεν συνέβη και στη συνέχεια και από την αποστολή δεν λάβαμε κάποια ε, απάντηση. Ε, έχετε δίκιο όμως ότι δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι όλο αυτό. χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονό ότι η αποστολή που θα μεταβεί ε, συντόμως ε, στην Μολδαβία ε, είναι διατεθειμένη στο πλαίσιο της προετοιμασίας, της προετοιμασίας για το ταξίδι να συζητήσει για να προετοιμαστεί πάνω σε αυτό ε, χαιρόμαστε δηλαδή και για όλο αυτό και είμαστε ευγνώμονες για την, ευγνώμονες για την προσφορά σας και θα σας υποστηρίξουμε σε αυτό. Κάτι το οποίο ε, ανέφερα ε, όσον αφορά το σκάνδαλο του ενός δισεκατομμυρίου. Ε, η κυβέρνηση θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει μόνη της αυτό. Κάτι το οποίο βοηθάει είναι το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, το οποίο αποτελεί ε, διασφάλιση ποιότητας ε, για την διαχείριση χρημάτων και πόρων στην χώρα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολλά όσον αφορά την διαφθορά. Με την κυβέρνηση της Μολδαβία. έχουμε συζητήσει πολύ για αυτό. Κάθε συνάντηση που έχουμε στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης το, χρησιμοποιούμε κάθε ευκαιρία για να το κάνουμε αυτό και έχουμε καλά αποτελέσματα. Τώρα το ερώτημα ε, σχετικά με το τι μπορούμε να κάνουμε. Ε, το δικό σας τελευταίο ερώτημα κυρία Πρόεδρε. Πράγματι δεν ε, έχουμε μια ισχυρή ε, θέση. Ναι, κάποιες από τις ε, δεσμεύσεις είναι νόμιμες διότι έχουμε ένα, ε, μια συμφωνία σύνδεσης όμως, όμως σε μια τέτοια περίπτωση μπορούμε να ξεκινήσουμε έναν κριτικό διάλογο, κάτι το οποίο κάνουμε όμως όπως προανέφερα θα θέλουμε να επικεντρωθούμε στην ε, οικονομική μας συνεργασία σε συγκεκριμένα ε, προγράμματα τα οποία ε, βοηθούν τους πολίτες εκτός από αυτά τα οποία συμφωνήθηκαν και θα πρέπει να τα συνεχίσουμε γιατί ήταν δική μας δέσμευση. Αυτό δεν αφορά τις δράσεις του 16 και έπειτα Έχουμε λοιπόν το μίσο που πιστεύουμε ότι μπορεί να υπάρξει ε, μια ε, καλύτερη ε, συνεργασία όπως είναι για παράδειγμα η συνδεσιμότητα, η εκπαίδευση. Η ικανότητά μας λοιπόν να ελέγχουμε και ε, να ε, δίνουμε μεγαλύτερη, να απαιτούμε μεγαλύτερη λογοδεσία για αυτά τα προγράμματα είναι μεγαλύτερη. Αυτό λοιπόν σκοπεύουμε να κάνουμε. Συμφωνώ λοιπόν ότι είναι πολύ σοβαρό για να το αγνοήσουμε και να το ξεχάσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να ε, συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε αυτό μέσω των αποστολών μας αλλά και σε άλλα φόρουμ όπως είναι η επερχόμενη επίσκεψη της αποστολής από τη Μολδαβία ε, δεν είμαι σίγουρος όμως ότι θα δούμε οποιασδήποτε αποδείξεις ε, με βάση ε, που αφορούν τις κατηγορίες του Προέδρου. Ευχαριστώ πολύ. Τότε θα πρότεινα λοιπόν να μας δώσετε μια λίστα με όλες τις αξιολογήσεις των τελευταίων χρόνων αλλά και τις προβλεπόμενες αξιολογήσεις τις οποίες θα τις εξετάσουμε λεπτομερώς εμείς ε, και στη συνέχεια ε, πιστεύω ότι εφ' εξής ε, θα παρακολουθούμε στενά. Ευχαριστούμε λοιπόν και εσάς που θα μας ενημερώσετε για όλες τις συναντήσεις που θα έχετε με ε, εισαγγελίες, με κοινωνίε των πολιτών ε, ε, και θα ήμασταν ευγνώμονες για οποιοδήποτε περαιτέρω πληροφορίες και για την ώρα θα θέλαμε να έχουμε μία δράση διότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε καθότι έρχεται σε αντίθεση με οτιδήποτε κάνουμε καθημερινά εδώ μέσα και με προσβάλλει προσωπικά διότι ε, θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να ε, ξαφνικά θα πρέπει να δικαιολογηθούμε για την δήλωση να δικαιολογηθούμε για το γεγονός ότι αγνοήσαμε τη δήλωση ενός προέδρου λέγοντας ότι παίζει ή δεν το εννοεί έτσι αυτή είναι η άποψή μου λοιπόν και αυτό θα πράξουμε. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τις περαιτέρω πληροφορίες που μας δώσατε. Ε, και όσον αφορά την υποστήριξη του προϋπολογισμού και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα διότι γύρεται το ερώτημα ε, διότι θα θέλαμε και πληροφορίες σχετικά με το πώς εξετάζεται η εφαρμογή του προϋπολογισμού και ε, θα θέλουμε λοιπόν ότι η επόμενη επίσκεψη της ε, Μολδαβίας ε, να μας ενημερώσετε πότε θα γίνει για να μπορέσουμε και εμείς να προσκαλέσουμε τον επικεφαλής της αποστολής διότι θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι να στείλουμε ένα σήμα ότι ε, δεν είμαστε οι ε, ε, τελευταίοι λύθοι του πλανήτη που ανέχονται το οτιδήποτε υπάρχουν ε, άλλες ε, προτάσεις ε, για βήματα τα οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε. Σας παρακολουθούμε, μην μας ξεχάσετε, μας είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης και μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 8 το οποίο αφορά το ταξίδι μας στην Ιορδανία και τον Λίβανο το Σεπτέμβριο του 2016. Πέρασε καιρός μέχρι ότου να ασχοληθούμε με την συγκεκριμένη επίσκεψη. Αρχικά πήγαμε ε, στο Λίβανο και στη συνέχεια στην Ιορδανία. Ήταν ένα ενδιαφέρον ταξίδι το οποίο επικεντρώθηκε ε, στην, ε, στα μέσα της ε, του Γραφείου Αραϊκής ε, και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, ένα ε, γραφείο το οποίο εργάζεται εδώ και 25 χρόνια περίπου. Έχουμε να κάνουμε με έναν τεράστιο αριθμό ανθρώπων Έχουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο τσουνάμι ανθρώπων οι οποίοι ε, θεωρούνται ε, πρόσφυγες ε, και έχουμε να κάνουμε όλες αυτές τις συνέπειες. Με εξέπληξη ιδιαίτερο το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν σε σπίτια τα οποία ονομάζονται καταφύγια τα σπίτια αυτά όταν υπάρχουν προβλήματα ε, ε, τότε κάποιος άλλος θα πρέπει να τα επισκευάσει ε, αυτό το οποίο ε, με ξένησε ε, είναι ότι υπάρχει μια ότι οι άνθρωποι δεν έχουν την ευθύνη του μέλλοντός τους. Αυτό με συγκίνησε περισσότερο και το ερώτημα ε, που τίθεται είναι εάν η ε, ε, ανθρωπιστική βοήθεια που δίνεται έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να χάνουν τη δυνατότητα να καθορίσουν το μέλλον τους δεχθήκαμε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μας είπαν ότι τα χρήματα αυτά δεν επαρκούν, ε, είδαμε την ανεργία, είδαμε ότι στον ε, Λίβανο οι πρόσφυγες αντιμετωπίζονται χειρότερα από ό,τι στην Ιορδανία. ότι το 57% του προϋπολογισμού του Γραφείου Αρρωγής του ΟΗΕ ε, δίνεται ε, και ότι ε, υπάρχει ένας παγκόσμιος διεθνής συντονισμός για την αντιμετώπιση της διαμάχης Είδαμε επίσης ότι τα κράτη-μέλη εργάζονται κατά τόπους εκεί πέρα και προσπαθούν να απαλύνουν τον πόνο Στη ε, είδαμε ότι ε, στον Λίβανο ε, υπάρχει η δυνατότητα άσκησης 70 επαγγελμάτων όπως είναι οι γιατροί οι οποίοι όμως επιτρέπεται μονάχα να θαλπορούν τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες θα πρέπει λοιπόν να γίνει κάτι για όλο αυτό στην Ιορδανία τώρα επισκεφθήκαμε 10 ε, ε, στρατόπεδο συνόλικα, βρεθήκαμε και πολύ κοντά στα σύνορα με τη Συρία. Ε, προσπαθήσαμε να κινηθούμε τριγύρω για να συζητήσουμε με τους πρόσφυγες και είδαμε ότι υπάρχουν τυπικά προβλήματα όπου έχουμε ανθρώπους που έρχονται απ' έξω και θέλουν να κάνουν κάτι καλό. Είδαμε ότι τα σπίτια στα στρατόπεδα αυτά δεν έχουν τουαλέτες ή ότι ε, πολλοί άνθρωποι ε, χρησιμοποιούν μια κοινή τουαλέτα με αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να μην τολμούν το βράδυ ε, να βγουν έξω με αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη περιοχή του σπιτιού να χρησιμοποιείται για αυτό το σκοπό, διότι δεν υπάρχει φωτισμός για να πάνε στην κοινή τουαλέτα οι γυναίκε. κάτι τέτοιο δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ήταν για μένα απαράδεκτο το γεγονό ότι δεν υπάρχει κανένας ο οποίος ε, μπορεί να διορθώσει ε, τέτοια ε, λάθη. Προσωπικά το βρήκα απίστευτα λυπηρό. Ήταν όμως μια πολύ καλή προετοιμασία και για την επίσκεψη στα, στα κάμψη της Τουρκίας τώρα τι θα γίνει μελλοντικά με όλα αυτά τα ε, παλιά ε, στρατόπεδα στην Ιορδανία αλλά και στο Λίβανο. Ε, γύρεται συνεχώς αυτό το ερώτημα σχετικά με το αυτό αν όλα αυτά θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο διαβίωσης για τους πρόσφυγες ή αν τώρα θα πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια για ενσωμάτωση των ανθρώπων αυτών στην κοινωνία. Στην Ιορδανία ε, ο κύριος ε, Τσέλερ ε, θα παραδώσει την γραπτή έκθεση και η κυρία Κνίτσικ μπορείτε να μιλήσετε στα Ιταλικά, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ναι, προτιμώ πάντα να μιλάω Ιταλικά, είναι πολύ πιο εύκολο για μένα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εσάς αλλά και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτήν την αποστολή, η οποία πρέπει να πω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί πραγματικά μας έδωσε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτούς τους κατακλυσμούς συγγνώμη, καταβλισμούς και να καταλάβουμε πόσο περίπλοκη είναι η κατάσταση. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν ε, γιατί ε, πραγματικά όλοι είχαμε πολύ επικοδομητικό πνεύμα. Προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τα μάτια μας, να δούμε ακριβώς ε, τι συνέβαινε και ε, ακριβώς να μεταφέρουμε τα τεκτενόμενα έτσι ώστε καλύτερα να προετοιμάσουμε την ευρωπαϊκή παρέμβαση. Η κατάσταση είναι δραματική όπως τα είπατε όσον αφορά τις υγειονομικές συνθήκες τις συνθήκες διαβίωσης, όσον αφορά τα δικαιώματα, όλα αυτά που είδαμε στους καταβλισμούς των προσφύγων και στο Λιβανό και στην ε, Ιορδανία είναι ακριβώς όπως τα περιγράψατε. Εγώ θεωρώ ότι η κατάσταση στην Ιορδανία και νομίζω ότι συμμερίζονται όλη την άποψη ε, ε, αυτή, είναι καλύτερη η κατάσταση από ό,τι στο Λίβανο και ίσως τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα είναι αυτά τα οποία αφορούν την εκπαίδευση και την ε, διδασκαλία γιατί πραγματικά ε, δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ε, μετά από όλα αυτά που είδαμε, ε, πραγματικά έχω την εντύπωση ότι τα πιο αποτελεσματικά είναι τα προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά επίσης είναι τα προγράμματα κατάρτισης και προετοιμασίας ε, σε κάποιο επάγγελμα. Επίσης διαπιστώσαμε ότι στο Λίβανο υπάρχει και ένα πρόβλημα συμβίωσης των Παλαιστινίων προσφύγων και των Σύρων προσφύγων, γιατί η πολιτική κατάσταση είναι ήδη περίπλοκη, το πολιτικό πλαίσιο ήδη περίπλοκο και μπορεί να περιπληκθεί ακόμα περισσότερο. Διαπιστώσαμε επίσης ε, ότι οι συνθήκες συμβίωσης και διαβίωσης είναι πάρα πολύ ε, ε, έντονοι και βεβαίως εδώ ελοχεύει και ο κίνδυνος ρίζοσπαστικοποίησης. Ε, η κατάσταση και στις δύο χώρες ε, είναι δύσκολη όσον αφορά τα οικονομικά. Ε, μιλήσατε ήδη και αναφέρατε το υψηλό ποσοστό ανεργίας, την δυσκολία ένταξης των προσφύγων ε, στις δύο αυτές χώρες. Περίπλοκα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα δούμε με προσοχή και να τα αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα. Η οικονομική κατάσταση των δύο χωρών είναι αυτή που είναι ε, βεβαίως ε, διαπιστώσαμε ότι είναι πολλές οι προσπάθειες που καταβάλλονται από τις ε, τοπικές ε, και περιφερειακές αρχές αλλά τα προβλήματα είναι εκεί. Υπάρχουν υψηλό ποσοστό ανεργίας, αύξηση του δημοσίου χρέους στις δύο χώρες που κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Προβλήματα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, κυρίως σε σχέση με αυτό που είπατε για τα παιδιά και τις γυναίκες. Επομένως, παρέμβαση, υποστήριξη που μπορούμε να κάνουμε εμείς μέσα από τα προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται και η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την Ανακούφιση και, και τα έργα, η UNRWA ε, θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένες ε, και οπωσδήποτε στήριξη και μέσα, του ε, από το Ευρωπαϊκό Όργανο Γειτονίας. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε πέρα από την πολύ θετική αξιολόγηση εργασίας που γίνεται ε, είναι ότι οπωσδήποτε ε, πρέπει να υποστηρίξουμε ε, την κατάσταση γιατί η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη, οι συνθήκες στις χώρες είναι δύσκολες. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος διαφθοράς. Θα πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναμφίβολα πάντως, και αυτή είναι η αίσθηση που αποκόμισα εγώ, βάσει της εμπειρίας αυτής της αποστολής που ήταν πραγματικά πάρα πολύ βαριά και από ψυχολογική ε, άποψη γιατί είδαμε πράγματα τα οποία τα ακούμε, τα συζητάει, ε, τα συζητάει ο κόσμος αλλά πραγματικά ε, δεν ήταν δυνατόν να τα συνειδητοποιήσουμε πριν τα δούμε αυτούς τους τεράστιους καταβλισμούς ε, που απλώς ενισχύουν ακόμα περισσότερο την ε, βούλησή μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς έτσι ώστε να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζέλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, Κάτι που ε, πρόσεξα και εγώ εκεί πέρα είναι ότι όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης ε, στο ε, Λίβανο που έχουν οι Παλαιστίνοι δεν αποτελεί θαύμα, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, το, ότι η Χεσμολά δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα να βρει στρατιώτες διότι η Χεσμολά είναι ιδιαίτερα ενεργή εκεί πέρα, έχει την υποστήριξη του Ιράν με όπλα και ε, βλέποντας και σε περίπτωση που δεν αλλάξει τίποτα στο Λίβανο και στην Ιορδανία τότε σίγουρα θα υπάρχει, υπάρξει περαιτέρω ακρεοποίηση ε, και ε, βλέποντας τις τυχογραφίες στα σπίτια τότε όλα υποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί. Ε, πριν από 70 ε, χρόνια, το 48 ε, νομίζω, δημιουργήθηκε η UNRWA, η οποία όμως λαμβάνει χρηματοδότηση από την κυρίως, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρόλο που είναι οργάνωση του ΟΗΕ. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς είναι δυνατόν εμείς να σηκώνουμε το μεγαλύτερο βάρος της χρηματοδότησης, διότι πρόκειται για θεσμική χρηματοδότηση ε, και ε, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι. Τα ΟΗΕ θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του, διότι ε, η περαιτέρω χρηματοδότηση γίνεται από τις ΗΠΑ και κατά 10% από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι το ένα θέμα. Από την άλλη, οι άνθρωποι βρίσκονται εκεί σε τέταρτη-πέμπτη γενιά. Παρόλα αυτά θεωρούνται Παλαιστίνοι, παρόλο που ελάχιστοι εξ αυτών γεννήθηκαν στην Παλαιστίνη όμως ε, δεν βοηθούνται καθόλου για να υπάρξει ε, ενσωμάτωση ε, στις χώρες. Στην Ιορδανία τουλάχιστον έχουν το δικαίωμα να εργαστούν στο Λίβανο όμως δεν έχουν ούτε καν αυτό το δικαίωμα. Δηλαδή ναι μεν ε, εκπαιδεύονται ε, και καταρτίζονται, δεν έχουν καμία δυνατότητα στο Λίβανο όμως να εργαστούμε. δεν μιλάμε όμως για καταβλισμούς κάτι ακόμα, πρόκειται για γκέτο. Ε, πρόκειται για περιοχές πυκνοκατοικημένες, ε, έχουν γίνει ε, δρόμοι όπου υπάρχουν ερήπια, δεν είναι σπίτια αυτά και οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τη ζωή τους να χάνεται εκεί πέρα ε, και οποιαδήποτε δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα που γίνεται εκεί πέρα είναι μια παράνομη, είναι μια ανεπίσημη οικονομία ε, παράλληλα με αυτά τα γκέτο, δεν μπορεί να είναι ε, το μέλλον όλο αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε σοβαρά και άμεσα το πώς λοιπόν θα συζητήσουμε με τους υπευθύνους οι οποίοι δεν βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά στον ΟΗΕ και πώς θα συνεργαστούμε με αυτούς. Ε, η τελευταία ε, δήλωση τύπου την οποία συζήτησε, την οποία ε, έπεσε στα χέρια μου έδειξε ότι η χρηματοδοτικές ανάγκες αυτού του οργανισμού για να μπορεί να κάνει το μήνυμο του έργου της όσο πάνε και μειώνονται ε, τα ε, κράτη-μέλη εργάζονται πάνω σε ε, προγράμματα, κάτι το οποίο είναι σύνηθες, όμως αποτελούν απλά μια σταγόνα στην καυτή άμμο. Έχουμε δύο τομείς φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών ε, το δεύτερο λοιπόν ε, η αφορά τους ε, πρόσφυγες από την Συρία οι οποίοι έχουν πάει σε γειτονικέ χώρες και οι πόλεις αυτές και οι περιοχές αυτές αποτελούν ένα κίνδυνο διότι αποτελούν ε, μια μεγάλη ε, πλειοψηφία στις χώρες αυτές ε, και βλέποντας το πώς την προσπάθεια των πόλεων αυτών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα να ενσωματώσουν αυτούς τους ανθρώπους βλέπουμε ότι λάβανε 1,2 δις υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ε, από τη διεθνή κοινότητα ε, και εδώ έχουμε τη δεύτερη οργάνωση του ΟΗΕ το οποίο είναι η ύπατη για τους ε, πρόσφυγες όλα αυτά ανταγωνίζονται μεταξύ τους ε, σχετικά με το ποιος ε, θα λάβει τα μέσα για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του ε, και πάλι εδώ βοηθάει ιδιαίτερως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ερώτημά που είναι τι ακριβώς κάνει ο ΙΕ ο οποίος κανονικά είναι υπεύθυνο για, αυτές τις, για αυτούς τους οργανισμούς και αν λοιπόν εμείς είμαστε ε, βασικοί χρηματοδότες αυτών των ε, οργανισμών τότε δεν θα έλεγα ότι δεν κάνουν ε, σωστή δουλειά όμως δεν θα τολμούσα να κάνω κάτι τέτοιο όμως θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς μπορούν να καταρτιστούν καλύτερα ε, αυτά τα οποία είπε η Πρόεδρος είναι ολόσωστα ε, και επίσης πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους ε, για ζητήματα αυτοβοήθειας, για το πώς μπορούν να εκπαιδευτούν, να καταρτιστούν ηλεκτρολόγοι ή άλλα τέτοια επαγγέλματα και το πώς μπορούν να χρησιμοποιούν τα υλικά εκεί πέρα για να δημιουργήσουν σωστές περιοχές και να μην ζουν μέσα σε έναν σωρό από σκουπίδια, αρουραίος και ερήπια όπου οι νέοι δεν δεν έχουν καμία προοπτική ε, για το μέλλον και γίνονται εύκολη ε, λία για ε, ε ακραίες οργανώσεις που στο μεταξύ έχουν επεκταθεί ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά όλα είναι τα προβλήματα τα οποία δεν θα πρέπει να τα σπρώχνουμε κάτω από το πατάκι. Ευχαριστώ πολύ. Ε, όσον αφορά ε, τους ηλεκτρολόγους αυτή είναι η σωστή ε, λέξη διότι υπάρχουν κάθε χρόνο εκατοντάδες νεκροί από ηλεκτροπληξίες. Η κυρία ο κύριος Παπαχέβριας Ευχαριστώ πολύ Κυρία Πρόεδρα Ευχαριστώ πολύ για τα όσα μας αναφέρατε. Θα τα λάβουμε όλα αυτά πολύ σοβαρά υπόψη. Βεβαίως, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Και ο κύριος Τσέλερ πολύ σωστά ανέφερε ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες προσφύγων. Έχουμε πολλές γενναίες Παλαιστινίων που μένουν, διαμένουν στην Παλαιστίνη και στο Λίβανο. Έχουμε Σύρους πρόσφυγες ή και Σύρους δεν είναι όλοι πρόσφυγες. Γι' αυτό υπάρχει σύγχυση ακόμα και για τα αριθμητικά στοιχεία. Η τελευταία απογραφή αναφέρει ότι ο πληθυσμό είναι 1,3 εκατομμύρια, αλλά μόνο η μισή από αυτού είναι πρόσφυγε. Όμω υπάρχει τεράστιο άχθο ε, και πίεση και στι δύο αυτέ χώρε. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε και θα κάνουμε ό,τι πρέπει από το χέρι μα για να του βοηθήσουμε αξιοποιώντας ε, διμερή ε, χρηματοδότηση, η e ΕΝΑΗ, και το πιο σημαντικό είναι το καταπίστευμα Μαντάντ για τη Συρία. Και συνεργαζόμαστε με όλους τους εταίρους που έχουμε επιτόπου. Ε, ο οργανισμός UNRWA, όντως, η ΥΠΑΤΗ Αρμοστία για τους πρόσφυγες, ιδίως στην Ιορδανία. Το είδατε και μόνοι σας. Αλλά και εγώ επισκέφθηκα τον ίδιο καταβλισμό στην Ιορδανία μερικές εβδομάδες πριν από εσά. Υπάρχουν σημαντικέ διαφορές ε, στην ε, κατάσταση εκεί. Οι καταβλισμοί στην Ιορδανία είναι πολύ μεγαλύτεροι και πολύ καλύτερα οργανωμένοι. Ενώ στο Λίβανο οι περισσότεροι από του πρόσφυγε ε, διαμένουν σε μικρές, μικρούς καταβλισμούς, μικρές κατασκηνώσεις αν θέλετε, που βρίσκονται διάσπαρτοι ε, σε όλη την επικράτεια. Νομίζω και στην ίδια την ε, διάδα ΒΕΚΑ είναι χιλιάδες. Τώρα, πιο συγκεκριμένα κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτον, για την συνεργασία μας με την ΟΝΡΟΑ, τον οργανισμό του ΟΗΕ, που νομίζω είναι και ε, ο παλαιότερος οργανισμός του ΟΗΕ. Εδώ και 70 χρόνια εφίσταται. Είμαστε ως Ευρωπαϊκή Ένωση ο πιο προβλέψιμος ε, χορηγός, δωρητής προς ε, τον ε, οργανισμό και αυτό θα συνεχιστεί. Συνήθως υιοθετούμε μια κοινή διακήρυξη μαζί τους, ούτως ώστε να προβλέπετε χρηματοδότηση, να μπορούν και αυτοί να κάνουν το μακροχρόνιο σχεδιασμό τους και έχουμε προετοιμάσει μια νέα διακήρυξη για την συγγνώμη, περίοδο 2014-2020 που θα πρέπει ακόμα να υιοθετηθεί επισήμω. Όμω ε, παραμένουμε και διατηρούμε ένα σταθερό επίπεδο χρηματοδότηση των 82 εκατομμυρίων ευρώ κατά έτο. Πράγματι, αυτό το ποσό δεν επαρκεί. Παρεμπιπτόντω, να ξεκαθαρίσω την κατάστασή μα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μέλο ε, εδώ έχουμε καθεστώς παρατηρητή. Βεβαίως όλα τα μέλη μας είναι μέλη του ΟΗΕ. Ναι, αυτό είναι ένα εσωτερικό πρόβλημα πολλών οργανισμών, ιδίως της ΥΠΑ της Αρμοστίας για τους πρόσφυγες. Σε ένα βαθμό και άλλοι. ουσιαστικά έρχονται όλοι αυτοί οι οργανισμοί αντιμετώπιοι με ένα τεράστιο πρόβλημα χρηματοδότηση. Και ξέρετε ότι το κενό στον προπολογισμό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένε αποφάσει από ορισμένα κράτη-μέλη του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Εμεί όμω θέλουμε να είμαστε προβλέψιμο εταίρο και προ αυτήν την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε να κινούμεθα. Έχουμε σχετική, σχε, τέτοιες συστηματικές ανταλλαγές πληροφοριών με τον Ούνουρα και με τον κύριο Κρένμπουλ, ε, επικεφαλής ε, του οργανισμού αυτή τη στιγμή. Και σαφώς και, και αυτοί επιτελούν το σκοπό τους. Το ίδιο ισχύει και για την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες. Τρέχουν όλες τις υποδομές, όλους τους καταβλισμούς στην Ιορδανία. Και μάλιστα είναι και πολύ ποιοτική η δουλειά που κάνουν. σωστά παρατηρήσατε ότι δεν πρέπει να ενθαρρύνουμε ή μάλλον δεν πρέπει να αφαιρούμε την αξιοπρέπεια αυτών των προσφύγων, να τους βοηθήσουμε αντιθέτως ε, να έχουν μια κανονική ζωή στο βαθμό του δυνατού και δεδομένων των συνθήκων. Δεν καλύπτουμε λοιπόν τι καθημερινέ του ανάγκε επιβίωσης, αλλά επενδύουμε και στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική κατάρτιση και τεχνική κατάρτιση, ιδίω στο Λίβανο, αλλά και ευρύτερα, αν δείτε την κατάσταση, τι μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε την καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασία. Πριν έρθω εδώ σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, ε, ο Επίτροπος Χάν είχε διοργανώσει μια εκδήλωση σχετικά με τι επενδύσει εκεί και εξαιτία του συμφώνου που ε, υπογράψαμε με την Ιορδανία πέρυσι, του δώσαμε πολύ καλύτερες ε, συνθήκες πρόσβασης στην Ευρωπαϊκή Αγορά εργασία. Αλλάξαμε αυτού τους κανόνες προέλευση, να μην σας κουράσω τώρα με τις λεπτομέρειες, αλλά οι ίδιοι οι Ιορδανοί που ε, παρευρέθησαν εκεί είπαν και από την κυβέρνηση και από τον ιδιωτικό τομέα ότι αν ίσχυαν αυτοί οι κανόνε προέλευση, για παράδειγμα στον τομέα τη κλωστοϊφαντουργία ή στο πλαστικό, αυτό θα δημιουργούσε πάνω από 200.000 θέσει εργασία. Και ο όρο που είχε τεθεί ήταν ότι θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν τον αριθμό σημαντικό αριθμό προσφύγων. Έχουν ειδικέ οικονομικέ ζώνε λοιπόν και στην πρώτη φάση περιμένουμε ε, μια αναλογία, ένα ποσοστό 15% προσφύγων, το οποίο μετά θα πρέπει να γίνει 35%. Θα έχει λοιπόν θετικά αποτελέσματα εν καιρό. Αυτό όμως θα βοηθήσει πολύ τις δυνατότητες ε, απασχόλησης ε, των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Υπήρχε το θέμα των αδειών παραμονής και εργασίας. Στην Ιορδανία τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα από ότι στο Λίβανο υπήρξαν κάποιες θετικές εξελίξεις και εξακολουθούμε να ασκούμε πιέσει ε, στην κυβέρνηση. Για παράδειγμα, οι Παλαιστίνοι πρόσφυγε από τη Συρία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Λίβανο ε, έχουν ε, απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολή τέλους για να πάρουν τέτοια άδεια. Για το Λίβανο πιο συγκεκριμένα τώρα. Έχουμε συμφωνία σύνδεσης με αυτή τη χώρα. Όσο εκ τούτου, τα γεωργικά και μηχανικά προϊόντα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση άνευ ε, δασμών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν ακόμα προβλήματα σε ό,τι αφορά τα φυτογενομικά πρότυπα και την έλλειψη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο και για το εμπόριο, βεβαίω και για τι δυνατότητε απασχόληση και των ε, ίδιων των υπηκών του Λιβάνου και για του πρόσφυγε ε, που βρίσκονται εκεί. Τι να κάνουμε τώρα για το άχθο. Θέλουμε να επενδύσουμε όσο μπορούμε στις ε, συνθήκες διαβίωσης, στην τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση εδώ νομίζω ότι έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αυτό αναγνωρίζεται και από τις ε, δύο χώρες. Θετική εξέλιξη είχαμε και για το Λίβανο, γιατί παλαιότερα δεν είχαμε ούτε πρόεδρο, ούτε κυβέρνηση. Τώρα υπάρχει και πρόεδρος και κυβέρνηση. Πολύ πιο εύκολα και δομημένα μπορούμε να στηρίξουμε αυτή τη σχέση. Δεν είχε καν προπολογισμό για 8 χρόνια αυτή η χώρα. Απλώς ε, υπήρξε, υπήρχε μια μεταφορά του προηγούμενου προπολογισμού στην ένα rollover για την επόμενη χρονιά. Και μα επέκριναν γιατί δεν του στηρίζαμε αρκετά. Αλλά πώ μπορούμε να δώσουμε τη στήριξή μα όταν δεν υπάρχει προπολογισμό. Την περασμένη φορά ήμουν εκεί με μια ομάδα ε, πρεσβευτών και το ανέφερα πολύ ομά στον Πρωθυπουργό. Έχουν αλλάξει τώρα τα πράγματα. Και αυτό διευκολύνει τα πράγματα και για εμάς. Όταν όμως μιλούμε για καταμερισμό του άχθους και μιλήσετε για την δέσμευση και εμπλοκή των κρατών μελών που είναι θεμελιώδης σημασία και η συμμετοχή των κρατών μελών επί τόπου για ε, την εφαρμογή των σχεδίων και για, την, για τον κοινό πραγματισμό όλα βαίνουν καλώς. Όμω, η άλλη όψη του νομίσματο είναι η επανακατανομή των προσφύγων. Και ξέρετε ότι αυτή ε, η ιστορία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τους ηγέτες μας για ε, τα προγράμματα ανακατανομής δεν έχουν ακόμα εφαρμοστεί επαρκώς. Τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τέλη Απριλίου ανέφεραν ότι περίπου 18.000 πρόσφυγες έχουν ε, επανακατασταθεί από τον ε, συνολικό αριθμό των 160.000. Συνεχώς λοιπόν υπενθυμίζουμε στα κρατημέλη αυτό το γεγονός γιατί θα συμβάλλει τα μάλλα στην ελάφρυνση του άχθους για αυτές τις δύο χώρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι, δεν μπορούμε να ρίξουμε στην Κομισιόν την επίλυση ε, ε, διεθνών προβλημάτων, όμως, όμως ε, θα ε, κάνουμε μια στατιστική ε, ε, και θα ασχολούμαστε με καταπλησμούς τους οποίους χρηματοδοτούμε εδώ και 50-60 χρόνια εργαζόμαστε πάνω σε αυτό διότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι όμως η κατάσταση έχει ως έχει και σίγουρα θα ε, συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα και περνάμε ε, στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξη, το οποίο αφορά το ταξίδι που κάναμε στην Τουρκία από 2 μέχρι 4 Νοεμβρίου το 2016 όταν ε, ο ε, πρεσβεστής ε, της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι χαίρεται που έρχεται η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Μπορούμε να καταλάβουμε πόσο σοβαρή η κατάσταση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αποστολή αλλά και τις δύο αποστολές στην Ιορδανία και το Λίβανο αλλά και όσον αφορά την τουρκική αποστολή που μας συνόδευσε ε, διανύσαμε με εκατοντάδες χιλιόμετρα ε, με το λεωφορείο ε, και είχαμε σημαντικές συζητήσεις με την τουρκική πλευρά ήταν ενδιαφέρον λοιπόν ε, και σημαντικό ε, να δούμε το γεγονός ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έκανε ένα μεγάλο λάθος άμα σταματούσε τις συζητήσεις για την ένταξη. Γι' αυτό το λόγο και εγώ και εδώ και στην Γερμανία έχω υποστηρίξει να μην σταματήσουμε τη συμφωνία για τους πρόσφυγες αλλά ούτε και να σταματήσουμε τις ενταξιακές συζητήσεις διότι άμα δούμε την πραγματικότητα κατά τόπους και αν συζητήσουμε με τους ανθρώπους εκεί πέρα τότε ε, συνειδητοποιούμε ότι ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, εκπροσώπους που δεν έχουν τη διάθεση να συζητήσουμε μαζί τους, οπότε μπορούμε να φανταστούμε να, συζητήσουμε μαζί μας, οπότε μπορούμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η κατάσταση αν δεν υπήρχε, ε, υπήρχαν αυτά τα εργαλεία μας. Ε, το 2005 ε, λοιπόν ε, κύριε Ζάλλερ εμείς ψηφίσαμε ε, για τη συνέχιση των συζητήσεων για την ένταξη. Είδαμε λοιπόν ε, συζητήσαμε αποκλειστικά με τη... για τη συμφωνία ε, που αφορά τα 3 δισεκατομμύρια για τους ε, πρόσφυγες αλλά και, την... και τις προενταξιακές ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Είδαμε επίσης ότι η Τουρκία δεν ενδιαφέρεται πλέον για αυτές τις ενισχύσεις τα χρήματα αυτά είναι διαθέσιμα όμως δεν τα χρησιμοποιεί η Τουρκία ε, και ε, όλα αυτά έχουν να κάνουν ε, με τη δημοκρατία, με τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης όλα αυτά μετά το πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 είδαμε λοιπόν ότι με το, το πραξικόπημα άλλαξε η διάθεση στην Τουρκία και βλέπουμε ότι αλλάζει ακόμα πιο πολύ η διάθεση των πολιτών για μέτρα ιδιαίτερα μετά και το δημοψήφισμα ε, όσον αφορά τους ε, δημοσίους υπαλλήλους ε, οι οποίοι μέχρι στιγμής ήταν υπεύθυνοι για τα ευρωπαϊκά κονδύλια, πώς εξ αυτών εργάζονται και ποιοι όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τορκική πλευρά απουσίαζε όλο και κάποιος εταίρος, υπήρχε εμπόδιο από την πλευρά της Άγκυρας, όμως είδαμε ότι υπήρχαν χάσματα και έχουμε καθυστερήσει τρεις με πέντε μήνες ε, το ερώτημα αυτό μας εκπλήξει το οποίο, ε, εκπλήσει το οποίο μπορείτε να το καταθέσετε και γραπτό. θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό είδαμε ότι Ε, τι σημαίνει το να είσαι ε, πρόσφυγας, ε, είδαμε καταβλισμούς, είδαμε τους ανθρώπους εκτός των καταβλισμών, συζητήσαμε μαζί τους, είδαμε πόσο δύσκολη είναι η οικονομική κατάσταση για τους πρόσφυγες εκεί πέρα και πόσο σημαντική είναι η συμφωνία με την Τουρκία για τους πρόσφυγες, διότι δεν, το θέμα δεν είναι να στέλνουμε πρόσφυγες πίσω όταν προσπαθούν να περάσουν το Μεσόγειο, αλλά να τους βοηθήσουμε και εκεί πέρα. είχαμε, μιλήσαμε με δύο ε, αντιπροέδρους της κυβέρνησης ε, και είχαμε σημαντικές ε, συζητήσεις οι οποίες βασίζονταν και επηρεάζονταν πολύ από την κατάσταση εκεί πέρα όπου μας δήλωσαν ότι νιώθουν εγκαταλελειμμένοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ε, κατάσταση βέβαια στην Τουρκία έχει ε, χειροτερεύσει και γι' αυτό το λόγο θα μας ενδιέφερε ένα update της κατάστασης εκεί πέρα. Ε, ο κύριος Τσέλερ ζήτησε το λόγο όσον αφορά τις συζητήσεις για την ένδειξη. Δεν ξέρω αν θα αποφέρουν κάτι, όμως σίγουρα θα πρέπει να συνεχιστούν διότι είναι κάτι αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Ε, το ερώτημα είναι όμως ε, ποια είναι η πορεία ε, που θα ακολουθήσουμε και με ποια κατεύθυνση θα γίνει όλο αυτό, διότι πολλές καταστάσεις αλλάζουν συνεχώς όπως ανέφερε η Πρόεδρος ή δεν έχουμε εταίρους με τους οποίους μπορούμε να συζητήσουμε. Λιγοστεύουν συνεχώς. Με εξέπληξη με εξέπληξε μία ε, δήλωση ενός ε, εκπροσώπου της ε, Κομισιόν σχετικά με την εκπαίδευση των δικαστών ο οποίος είπε ότι όλοι οι δικαστές οι οποίοι εκπαιδεύονται πάντως στο ευρωπαϊκό δίκαιο πλέον δεν εργάζονται. Οπότε ποια είναι τα συμπεράσματα. Δεν είναι άσχημο όλο αυτό, διότι θα έχουμε νέους αποφύτους από το Πανεπιστήμιο, οι οποίοι θα εργαστούν ως εισαγγελείς και δικαστές, τους οποίους θα μπορέσουμε εκ νέου να εκπαιδεύσουμε πάνω στο ευρωπαϊκό ε, δίκαιο από μηδενική βάση. Δεν ξέρω αν αυτό ε, είναι αισιοδοξία ή αν αποφέρει κάτι. Ε, το, έχω, ότι υπάρχουν προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται όπως για παρεδειγμα η κατασκευή ε, σιδηροδρόμων αρχικά αφορούσαν την σύνδεση με τα ε, διευρωπαϊκά δίκτυα. Ε, όλο αυτό όμως υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Ε, παρόλα αυτά θα πρέπει να συνεχιστούν να συνεχιστεί η χρηματοδότησή τους δεν ξέρω αν όλο αυτό θεωρείται προεταξιακή ενίσχυση. Μόνο το 15% των προσφύγων από τη Συρία βρίσκεται σε καταπλησμού Οι υπόλοιποι ε, προτίμησαν ε, να μην πάνε στους καταβλισμούς διότι έτσι δεν έχουν καμία επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, είναι αποκλεισμένοι ε, δεν έχουν καμία σχέση. Εμεί πήγαμε στον καταπλησμό μαρά, το οποίο θεωρείται και το καλύτερο, τα άλλα δεν μπορέσαμε να τα επισκεφθούμε. Στο μεταξύ γύρεται και ένα δεύτερο ε, πρόβλημα στην Τουρκία, το οποίο δεν συζητάται ανοιχτά, το οποίο η διαμάχη με τους Κούρδους είχε ως αποτέλεσμα 60 ε, χωριά στα νότιο-ανατολικά να καταστραφούν Έχουμε ε, δηλαδή περιοχές ε, με ισχυρό κουρδικό ε, στοιχείο. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν και, και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάπου θα πρέπει να μείνουν και δεν ξέρουμε αν αυτό θα χρηματοδοτηθεί από εμάς στο πλαίσιο της προσφυγικής βοήθειας ή αν θα το λύσει η Τουρκία από μόνη της. Ο κύριος από την Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σας δώσω μία ενημέρωση όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί πολλά συμβαίνουν τελευταία ε, στην Τουρκία. Τον τελευταίο μήνα ή μάλλον περισσότερο από την απόπειρα πραξικοπήματος ε, τον περασμένο Ιούλιο. Κάποια από τα μέτρα μετά την απόπειρα πραξικοπήματο ε, είναι πολύ σοβαρά σε ό,τι αφορά την, ε, το σεβασμό του κράτου δικαίου, των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων, της αντιμετώπιση των δημοσιογράφων. Πολλοί έχουν φυλακιστεί. Ο υψηλότερο αριθμός φυλακισμένων δημοσιογράφων στον κόσμο βάσει των οργανισμών παρακολούθησης. Αυτά αναφέρονται και στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που δημοσιεύθηκε πέρυσι. Και τα έχουμε ήδη διαβιβάσει και τα διαβιβάζουμε συστηματικά στις τουρκικέ αρχές. Μετά είχαμε το δημοψήφισμα, στο οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση απάντησε αμέσως και δημοσίως στηρίξαμε και τα πορίσματα ε, του ΟΣΑ ε, υπήρχαν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά ε, τις συμπεριφορές που παρατηρήθηκαν. Όμως όλα αυτά θα ε, αξιολογηθούν σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση τη Τουρκία ω υποψήφια προ ένταξη αλλά και ω μέλου του ΟΗΕ. Εμεί δεν έχουμε κατακρίνει την Τουρκία για το γεγονό ότι έχει αλλάξει και πλέον είναι ε, προεδρικό το σύστημα, αλλά για τι ε, άλλε διαδικασίε που τρέχουν σε αυτή τη χώρα. Υπήρξε μία επίγουσα συζήτηση πριν από μία εβδομάδα στο Κοινοβούλιο και ο Επίτροπος Χαν ε, παρευρέθη Ήταν μια πολύ ζωντανή συζήτηση και την περασμένη Παρασκευή και οι Υπουργοί Εξωτερικών ε, συζήτησαν την κατάσταση στην Τουρκία μετά το, το, συγγνώμη, το δημοψήφισμα ε, στο άτυπο συμβούλιο στη Μάλτα. Νομίζω ότι κανείς ή μάλλον τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα θέλουν να διατηρήσουν ένα διάβλο επικοινωνία με την Τουρκία Θέλουμε να συνεχιστούν οι επαφές μας. Γι' αυτό και συνεχώς θα αξιολογούμε την κατάσταση και στις επόμενες εβδομάδες. Γιατί η κατάσταση μεταβάλλεται συνεχώς. Όμως ε, δεν αποχωρούμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ο τουρκικός λαός πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο του διαλόγου μας καθώς και η οικονομική μας ε, συνεργασία θα συνεχιστεί, θέλουμε να επικεντρωθούμε πραγματικά στην κοινωνία των πολιτών και στις ε, θεμελιώδεις ελευθερίες. Γιατί αυτό είναι το κύριο μέλημα προς το παρόν. Κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, των διωγμών που ακολούθησαν την απόπειρα πραξικοπήματος. Τα τελευταία στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι πάνω από 96.000 δημόσιοι υπάλληλοι ε, απολύθηκαν σε όλους ε, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες. Σε ό,τι φορά τους ε, προτιμόμενους συνομιλητές μας, στο Υπουργείο Εξωτερικών περίπου 400, 383 πιο συγκεκριμένα, το Υπουργείο σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επηρεάστηκε τόσο πολύ, μόνο 20 υπάλληλοι απολύθηκαν. Επομένω, σε άλλα υπουργεία αυτό ήταν πολύ ε, περισσότερο. Ανησυχητικά όλα αυτά, όμω όλα εξαρτώνται από τον ε, τομέα συνεργασία. Σε άλλου τομεί είχαμε ε, μεγαλύτερε απώλειε από τι σε ορισμένου. Τώρα, για την συμφωνία με τους πρόσφυγες, για την συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας ε, είναι πολύ σημαντική. Όπως είπατε και εσείς, συμφωνώ ότι πρέπει να συνεχίσουμε την εφαρμογή της συμφωνίας. Η 15η έκθεση για την εφαρμογή της συμφωνίας με την Τουρκία και η πρώτη ετήσια έκθεση για τη διευκόλυνση για την Τουρκία δημοσιεύθηκαν και οι δύο στις 2 Απριλίου. Παρόλη την κατάσταση μπορούμε να πούμε ότι ε, είναι επιτυχής η εφαρμογή των, ε, της συμφωνίας. Έχουμε κάποια απτά αποτελέσματα, κυρίως ε, σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της οδούς της, της Ανατολικής Μεσογείου. 97% πτώση των αφήξεων στην Ελλάδα και 93% στην Ιταλία. Πολλοί βέβαια εξακολουθούν να χάνουν τη ζωή τους, όμως πολύ λιγότεροι σε σχέση με πριν. Μέχρι το Μάρτιο το 2016 οι, ετή, οι ημερήσεις αφήξεις υπερέβαιναν τους 107.000 ε, ε, ανθρώπους. Τώρα, κατά μέσο όρο έχουμε, πέσει στους 49.50 50 κάθε μέρα. Και πάλι πολλοί είναι δεδομένη της κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Αλλά είναι κάτι το διαχειρίσιμο. Και εμείς εμένουμε στις δεσμεύσεις μας πρέπει να δώσουμε τα εύσημα στις τουρκικές αρχές για τα όσα κάνουν. Και κάνουν πολλά, γιατί έχουν υποδεχθεί περίπου 3 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες οι Τούρκοι. Οπότε το κράτος έχει απομειστεί ένα τεράστιο βάρος και εμείς τους βοηθούμε μέσω της διευκόλυνσης για τους πρόσφυγες στην Τουρκία. Όπως αναφέρατε, 3 δις ευρώ έχουν ε, διοχετευτεί εκεί, 2,2 έχουν ε, ε, τύχη ε, πίστοση, ε, υπάρχουν συμβάσει δισεκατομμυρίων και όλα αυτά οδηγούν σε 700 εκατομμύρια σε πληρωμέ. Τώρα δεν θέλω να σα κουράσω. Τα περισσότερα έργα αφορούν ε, τις κοινοτικές υποδομές, την υγειονομική περίθαλψη και την παιδεία. Τα περισσότερα έχουν εφαρμοστεί μέσω των εταίρων μα, η τη αρμοστέ τη πρόσφυγε, UNICEF, Παγκόσμια Τράπεζα, οργανισμοί ορισμένων κρατών μελών, όπω η Γερμανική Αναπτυξιακή Τράπεζα KfW. Αλλά είχαμε και άμεσες επιδοτήσεις προς την ε, τουρκική κυβέρνηση και πολλές φορές λάβαμε επικρίσεις από εκπροσώπου ε, τη κυβέρνηση, ότι δεν του δίναμε αρκετή οικονομική στήριξη. Αυτό δεν ισχύει όμω. Είχαμε δύο ε, πολύ σημαντικές επιχορηγήσεις ε, εκατομμυρίων ευρώ για τα Υπουργεία ε, Υγείας και Παιδείας στην Τουρκία. Να αναφέρω επίσης, για λόγους διαφάνειας και κατόπιν πρωτοβουλίας του Επιτρόπου Έτιγκερ θα θέλαμε να προσκαλέσουμε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει ως παρατηρητής στις, ε, στη Διευθύνουσα Επιτροπή. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Ιούνιο και περιμένουμε το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει. Για τον ε, προτεξιακό διάλογο, την προτεξιακή ε, συνδρομή προς την Τουρκία, πρώτα απ' όλα εξετάζουμε την συνεχιζόμενη ε, βοήθεια και στήριξη υπό τα εργαλεία ΙΠΑ. Είχαμε δύο κύρια έργα, ε, το ένα συμπεριλάμβανε την κατάρτιση και τα σταματήσαμε. Παρακολουθούμε την κατάσταση και θα προβούμε σε ορισμένε ενέργειες αν αυτό είναι απαραίτητο και ε, υπάρχουν διατάξεις που προβλέπουν την επιβράβευση καλών επιδόσεων ή της περικοπής δαπανών αν τα πράγματα δεν βαίνουν ικανοποιητικώς. Αυτές ε, οι αξιολογήσεις θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Θέλουμε να επανεστιάσουμε τη συνεργασία μας ε, σε μεγαλύτερο βαθμό να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών. Μπορώ να σας δώσω και άλλα στοιχεία για το πώς ε, λειτουργεί η διευκόλυνση. Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας βεβαίως. Κάτι τελευταίο για τη συνεργασία μας με την Τουρκία. Οι εργασίες που γίνονται για τον εξυγχρονισμό της Τελωνιακής Ένωσης. Αυτό το έχει συζητήσει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο. Στα τέλη της περασμένης χρονιάς η Επιτροπή υιοθέτησε εντολή για την επικαιροποίηση της Τελωνιακής Ένωσης για να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, γιατί υπάρχει εδώ και 20 χρόνια, να συμπεριλαμβάνει για παράδειγμα υπηρεσίες, δημόσιους διαγωνισμούς, τη γεωργία. Τα ενδυνάμει, ωφέλη συγκεκριμένα για την Τουρκία είναι σημαντικά και το γνωρίζουν. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση στο Συμβούλιο, είναι εξαιρετικά πολιτικό το θέμα όπως ε, καταλαβαίνετε, όμως θεωρούμε ότι είναι κέρια σημασία και μπορεί να αποτελέσει τη βάση μιας ε, πραγματικής ε, σταθερής σχέσης, όποιες και αν είναι οι πολιτικές αποφάσεις που θα ληφθούν στο μέλλον. Το κύριο μήνυμα όμω είναι να συνεχίσουμε την, ε, τις επαφές, ε, τη συνεργασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριο Στέλλα. Έχω μονάχα ένα ερώτημα σχετικά με τα τρία δις ε, βοήθειας για τους πρόσφυγες προς την Τουρκία. Ε, το ένα δις ε, θα έρθει από ε, τον προϋπολογισμό της Ένωσης και άλλα δύο από τα κράτη-μέλη. Αν κατάλαβα σωστά βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τις πληρωμής κάτω του δισεκατομμυρίου μέχρι στιγμής τα κράτη-μέλη με βάση τις ευθύνες, τις τους έχουν δώσει αρκετά ποσά όμως στη συνέχεια θα κληθεί να δώσουν αυτά τα χρήματα. Κανονικά ε, θα έπρεπε ε, να έχουν λάβει τις αποφάσεις για τον, στο πλαίσιο του προπολογισμού τους για αυτό. Όλα είναι υποέλεγχο, ε, ναι έχουν πληρώσει, υπάρχει μια διαδικασία κατά την οποία τα κράτη-μέλη λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό πληρωμής το οποίο λαμβάνω εγώ προσωπικά ως επικεφαλής αυτής της Επιτροπής Διαχείρισης φυσικά διαρκεί ε, περισσότερο ώστε να δοθούν τα συγκεκριμένη ποσά όταν μιλάμε για μεγάλα ε, προγράμματα ε, όπως είναι για παράδειγμα νοσοκομεία, σχολεία. Αυτή τη στιγμή πέρσι συζητήσαμε με την Παγκόσμια Τράπεζα για να κατασκευάσουμε σχολεία για 15.000 ε, παιδιά από τη Συρία. Αυτό βέβαια ε, θα ε, διαρκέσει παραπάνω και γι' αυτό το λόγο και οι πληρωμές θα δοθούν αργότερα. Όμως όπως και να έχει τα ποσά έχουν διασφαλιστεί και αυτό διαφέρει από το Ταμείο για τη Συρία όπου τα κράτη-μέλη ακόμα δεν έχουν αποδώσει. Ευχαριστώ πολύ. Όπως υπόθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είχε ε, επιφυλάξεις όσον αφορά ε, τα σχολεία. λεγόταν να χρησιμοποιούνται τα τουρκικά σχολεία όπου το πρωί θα πηγαίνουν τα παιδιά της Τουρκία, τα τουρκαϊκά και στη συνέχεια τα παιδιά της Συρίας. Ναι, η πρώτη πρόταση είναι να, έχουμε, να είχαμε βάρδιες Υπήρχε όμως και έλλειψη ε, σε δασκάλους ε, διότι δεν υπήρχαν αρκετοί δάσκαλοι που να μιλούν αραβικά. Ε, υπάρχει όμως μετεκπαίδευση αυτών με τη βοήθεια τη δική μας αλλά και τους UNICEF όμως η κατασκευή σχολείων και αυτό είναι μια προτεραιότητά μας, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία συζητάμε με την Παγκόσμια Τράπεζα θα κατασκευαστούν 70 νέα ε, σχολεία για 15.000 παιδιά από τη Συρία. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ε, να σας ε, μιλήσω, να σας μεταφέρω τα λόγια μιας δασκάλας μουσικής από τη Συρία η οποία μας είπε ότι δεν υπάρχουν μουσικά όργανα και ότι θα ήταν καλό για τα παιδιά να έχουν μπορεί να σας ακούγεται ε, ασήμαντο όμως σκεφτόμενοι το πώς ζουν τα παιδιά εκεί πέρα τότε αυτά τα μέτρα ε, σίγουρα ε, θα ήταν κάτι καλό και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να σας το τονίσω Βρισκόμαστε λοιπόν και ε, στο, τελειώσαμε και με, αυτή την, ε, με αυτό το σημείο. Θα συναντηθούμε αύριο στις 10. Ε, στις 9 έχουμε την συνεδρίαση των, συνεδρια... των συντονιστών. Τα λέμε αύριο.